Uh, Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Απασχόλησης. Ανακοινώσεις πρώτα. Έχουμε όλες τις γλώσσες με εξαίρεση τα φιλανδικά, τα βουλγαρικά και τα κροατικά. Σημείο 2. Ε, τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις. Πρώτον είχαμε τον τρίτο τριμερή διάλογο για το ISS είναι μια έκθεση του κυρίου Μέσεριτς που έγινε στις 16 του μηνός αυτή η συνεδρίαση. Ε, έχει επιτευχθεί πρόοδο σε κάποια θέματα και μεταξύ αυτών στις κατεξιότηση και ε, εφαρμοστικές, εκτελεστικές ε, πράξεις. Επομένουν κάποιες λεπτομέρειες να λυθούν. Η επόμενη συνεδρίαση ε, διαλόγου θα γίνει στο Στρασβούργο στις 31 Μαΐου το πρωί. Σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους και, ε, ε, από μεταλλαξιογόνες ουσίες και καρκιογόνες στην εργασία. Πρώτος και δεύτερος τριμερής διάλογος διεξήχθησε. Κλοντ αυτό έγινε στις 17 και στις 23 Μαΐου. Όλα τα βασικά θέματα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων και επιτεύχθη κάποια πρόοδος. Στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί και θα οριστικοποιηθεί το θέμα αρχές Ιουνίου σε τεχνικό επίπεδο. Ε, απομένουν ακόμα κάποια εκκρεμή ζητήματα και μεταξύ αυτών το θέμα του ντίζελ το οποίο θα συζητηθεί στον τρίτο γύρο τριμερούς διαλόγου που θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου. Δεύτερον, τριμερής διαλογή για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Έχει γίνει και εκεί κάποια πρόοδος. Υπήρξαν διάφοροι γύροι ε, τριμερούς διαλόγου. Ωστόσο, απομένουν ακόμα πολλά ζητήματα για να είμαστε ειλικρινεί που πρέπει να λυθούν. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 5 Ιουνίου. Τούτο λεχθέντο λοιπόν των ανακοινώσεων θα συνεχίσουμε το σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη όπου καλωσορίζουμε θερμά τον κύριο Ντομπρόφσκης και την κυρία Τέισεν. Έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τους επιτρόπους είναι ένα, τμήμα του διαρθρωμένου διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δώσουμε πρώτα ε, το λόγο στον Αντιπρόεδρο, κύριο Ντομπρόψκης, για να κάνει μια εισαγωγή και μετά ε, στην Επίτροπο την κυρία Τάισεν. Και μετά θα ε, ανοίξει η συζήτηση για σχόλια, ερωτήσεις από πλευρά των Ευρωβουλευτών. Λοιπόν, παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Ντομπρόφσκης. You can start. Ε, Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, καταρχάς ευχαριστώ για την πρόσκληση στον δομημένο, συμμετοχή μου στο δομημένο διάλογο. Έχουμε ακόμα ένα χρόνο μέχρι τις ευρωεκλογέ. Και τότε θα κριθούμε για αυτά που πετύχαμε σε αυτή την θητεία. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να εστιαστούμε επί αποτελεσμάτων. Πρέπει να εντείνουμε τις πολιτικές προσπάθειες για να υπερκεραστούν τεχνικά εμπόδια ούτως ώστε οι εκκρεμότητες να διευθετηθούν. Θα αναφερθώ στο ευρύτερο κοινωνικονομικό πλαίσιο στο οποίο γίνονται εργασίε και το πώς ευρωπαϊκός Πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο που πρόσφατα προτάθηκε θα βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Το 2017 η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτύχθηκε με ταχύτερο ρυθμό μετά από μια δεκαετία για πρώτη φορά από το 2007 όλα τα κράτη-μέλη είδαν τις οικονομίες τους ε, να αναπτύσσονται και φέτος αναμένουμε ανάπτυξη του ΑΕΠ να παραμένει ψηλό σε ρυθμό στο 2,3%. Αυτές οι βελτιώσεις γίνονται αισθητέ στην αγορά εργασίας. Η απασχολημότητα τώρα είναι πιο ψηλή από ό,τι κατά την κρίση και το επίπεδο της ανεργίας έχει σχεδόν επιστρέψει στα επίπεδα του 2008. Μακροπρόθεσμη ανεργία και ανεργία των νέων μειώνονται τα δημοσιονομικά έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι επενδύσεις ανακάμπτουν. Ε, παραμένουν όμως ευάλωτα σημεία. Ε, ε, λοιπόν, έχουμε άτυπη μορφές εργασίας που είναι σε ψηλότερο ποσοστό από ό,τι πριν την κρίση. Η σύγκληση οικονομική-κοινωνική πρέπει να στηριχθεί μέσω επενδύσεων και σε ανθρωπινό κεφάλαιο να γίνουν διαθετικέ μεταρρυθμίσει, να έχουμε ποιοτικέ απασχόληση, να αυξηθεί η παραγωγικότητα και να αναπτυχθεί το πραγματικό εισόδημα και να υπάρχει μια υπεύθυνη φορολογική πολιτική, δημοσιονομική πολιτική. Γι' αυτό έχουμε διαδικασία ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, νέα πλαίσιο προσανατολισμού Ευρωπαϊκών Πυλών και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε ένα νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μετά τη στο Γκέτεμπορκ τον Νοέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια διακήρυξη και δραστηριοποιήθηκε για να δώσει ουσία στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, διτό ο στόχο, σύγκληση προ τα άνω και να προσαρμοστούμε στις ταχείες αλλαγές της κοινωνίας μας. Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής ε, προόδου, αλλά είναι κρίσιμο και για μελλοντική ανταγωνιστικότητα. Όπως γνωρίζετε, η εφαρμογή του πυλώνα, η υλοποίηση του πυλώνα είναι κοινή προσπάθεια πολιτική. Τα κράτη-μέλη και θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ενώσης, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα πρέπει να παίξουν το ρόλο τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει αυτά που πρέπει την πλευρά τη. Ήδη παρουσιάσαμε βασικέ πρωτοβουλίε, παραδείγματο χάρη για διαφάνεια και προβλέψιμο πλαίσιο στι εργασίε, πρόσβαση σε κοινωνική προστασία για όλου και πρόταση για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για το εργατικό δυναμικό και θα αναφερθεί εκτενέστερα η Επίτροπος η κυρία Τάισαν από αυτό. Όσον αφορά το θέμα αυτό, πέρα τη νομοθεσία του Ευρωπαϊκό Εξάμεινο παίζει μεγάλο ρόλο για τις μεταρρυθμίσεις και την προώθηση κοινωνικής και οικονομικής πρόοδου επιτόπου από, το, φέτος λαμβάνει υπόψη και τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων και τώρα δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες διότι θα συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο στις 28 Ιουνίου σε κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Η χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι πολύ κρίσιμη για την υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων και να προωθεί την ε, ανωδική σύγκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τι 2 Μαου το κολέγιο εθέτησε την πρότασή τη για το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα ακολουθηθεί από συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδοτούμενα, χρηματοδότησης την επόμενη εβδομάδα. Ακολουθούμε πραγματιστική προσέγγιση ανταποκρινόμενη στο νέο πολιτικό πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την απόσυση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε σχεδιάσει σαφέστερα, απλούστερα και πλέον ευέλικτα τον μελλοντικό προπολογισμό από ότι τον τωρινό έχει ισορροπία μεταξύ παραδοσιακών και νέων πολιτικών προτεραιοτήτων. Και τώρα θα ήθελα να εστιαστώ επί δύο νέων οπτικών γωνιών υποστήριξη της σύγκλησης και επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Προτείναμε καταρχάς ένα πρόγραμμα υποστήριξη μεταρρυθμίσεων 25 δις ευρώ που θα προσφέρει οικονομική και τεχνική υποστήριξη στις μεταρρυθμίσεις και σύγκληση μέσω σύγκληση τα κράτη-μέλη που είναι καθοδόν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης έχουμε νέο, νέα λειτουργία για στεδροποίηση των επενδύσεων και των οικονομικών. Οι επενδύσεις στηρίζονται μέσω δανείων με εγγύσεις από το Ευρωπαϊκό Προπολογισμό μέχρι 30 εκατομμύρια ευρώ και επίσης κάλυψη των ε, πληρωμών των τόκων. Θέλουμε να επενδύσουμε περαιτέρω στο ανθρώπινο δυναμικό. Για να γίνει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο ενιαίο μέσο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ με πάνω από 100 δις ευρώ πρικοδότηση ε, ε, θα ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό των χρηματοδοτήσεων στον τομέα το κοινωνικό και παρά περικοπέ στην πολιτική συνοχή, το μερίδιο του ESF Plus εντό τη πολιτική συνοχή αυξάνεται από 23 πάει στα 27%. Επίση, εστιαζόμεθα επί της χρήσεως, διπλασιάζοντας το Erasmus Sins στα 30 δις ευρώ, το Ευρωπαϊκό ελληνικό Σώμα αλληλεγγύη το 1,26 δις ευρώ και προσημείωση πόρων για την ανεργία των νέων εντός του esf σύν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο Ταμείο για Επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση με κοινωνική θηρίδα και για βελτίωση του Ταμείου Προσαρμογή και Παγκοσμιοποίηση τη Ευρωπαϊκή Ενώση. Αυξήσαμε το νοτοτόριο, απλουστεύσαμε τη λειτουργία του μέσου και επεκτείναμε το πεδίο καλύψεω για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι αναταραχέ στην, στην αγορά εργασία. Συνδυάζοντα τι μεταρρυθμίσει και νέα στήριξη χρηματοδοτήσεω, θα ξεπεράσουμε τον κατακαιρματισμό των εργαλείων για να μπορέσουμε να επενδύσουμε στι δεξιότητε των ανθρώπων και να προωθήσουμε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ε, για μία ακόμη φορά, Τώρα ήρθε η στιγμή να εστιαστούμε επί αποτελεσμάτων, ούτως ώστε το έργο μας και το νομοθετικό και το οικονομικό να συμφωνηθεί πριν τι επικοί μα ευρωεκλογέ και το τέλο τη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβασιστείτε στη Μαριάν και σε μένα για να σα ε, διευκολύνουμε στην επίτευξη των συμφωνιών. Και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Μαριάν τώρα. Thank you, ε, Ευχαριστώ, Βάλτη. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Αυτό είναι το κοινό μέλημα της Επιτροπής σα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε πετύχει ήδη ε, πολλά στριμερεί διαλόγους για το Europass, για την απόσπαση των εργαζομένων και δείχνει ότι όπου υπάρχει θέλω υπάρχει και ένα μπορώ. Ακόμα και σε θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα, πάρα πολύ πολιτικά. Θέλω να ευχαριστήσω τους ηγητές και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σκληρή δουλειά τους και την προσήλωση στα θέματα αυτά. Βέβαια δεν έχουν τελειώσει τα θέματα. Μέχρι το τέλος της θητείας έχουμε πολλή δουλειά. Να σας αναφέρω τις πρωτοβουλίες που συζητάει αυτό τον καιρό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον οι συνομοθέτες, ο συντονισμός ε, των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, αναθεώρηση των κανόνων. Θέλουν και τα τρία θεσμικά όργανα οπωσδήποτε να προχωρήσουν και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια κινητικότητα των εργαζομένων δίκαιη. Τον Ιούνιο θα αποφασίσει το Συμβούλιο για τα δύο κρεμή θέματα και προσεχώς θα αρχίσουν διοργανικές συνομιλίες έτσι ώστε να κλείσει στην παρούσα θητεία αυτό το θέμα. Συνέργειες απόλυτη προτεραιότητα είναι να αντιμετωπίσουμε την πρώτη βασική επαγγελματική ασθένεια που είναι επαγγελματικός καρκίνος, που είναι πραγματικός δολοφόνος ε, στην ε, ε, εργασία. Για τις καρκινογόνες ουσίες έχει γίνει μια προσπάθεια. Έγιναν οι πρώτες συνεδριάσεις την περασμένη εβδομάδα και χτες το βράδυ, αν δεν απατώμε, έγινε και άλλη συνεδρίαση με επιτυχία και μπορώ να το πω αυτό και με μεγάλη προσοχή ε, βλέπουμε τις προτάσεις σας για τις εκπομπές καυσαερίων ε, κινητήρων πετρελαιοκίνησης. εξετάζοντα πάντα τη διηγήμενη νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρήπανση και τα καυσαέρια. Υπάρχει και ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα. Με την κοινή δήλωση είναι κοινή μα προσπάθεια και αυτή. Κάναμε πρόσφατα μια δήλωση, αλλά θα πρέπει τώρα να επιταχύνουμε τους ρυθμούς. Να επιταχύνουμε αν θέλουμε να βρεθεί μια συμφωνία ακόμα υπό βουλγαρική προεδρία. Γνωρίζω ότι το Κοινοβούλιο ήδη έχει δείξει και προθυμία και ε, επιθυμία να συνεργαστούμε. Ελπίζω και το Συμβούλιο να ανταποκριθεί τώρα. Αυτό θα είναι προς όφελος ε, όλων των πολιτών που έχουν αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι 80 εκατομμύρια και με τις εταιρείες σε μια ε, εσωτερική αγορά κατακαιρματισμένη και με δυσκολίες. Για την πρόταση ε, για την ισορροπία επαγγελματικού ιδιωτικού βίου χαίρομαι που διατηρείτε ψηλά τη φιλοδοξία και εσείς στην πρότασή μας. Πρέπει να εγκριθεί ε, κατά την παρούσα θητεία αυτή η οδηγία ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για πολλούς Ευρωπαίους άνδρες και γυναίκες αλλά και για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα 370 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο χάνουμε ε, λόγω των ε, διακρίσεων με βάση το φύλλο και το χάσμα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το θέμα και πρέπει να κλείσει. Ε, διαφανής και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Αυτή η πρόταση έρχεται να ακολουθήσει τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και ανταποκρίνεται στην αύξηση της επισφαλούς εργασίας, όπως το είπατε και εσείς πρόσφατα στα ψηφίσματά σας. Το Συμβούλιο προσπαθεί να βρει μια κοινή θέση τον Ιούνιο και ελπίζω οι δύο συνομοθέτες να φροντίσουν αυτή η σημαντική πρωτοβουλία να εγκριθεί το πολύ μέχρι την άνοιξη του 2019. Οι τριμερείς ε, οργανισμοί τώρα γίνονται διαπραγματεύσεις για τον ιδρυτικό κανονισμό ε, ε, Eurofound και Σεντεφόπ. Ξέρω ότι εκτιμάτε το έργο των οργανισμών αυτών και γι' αυτό χρειάζεται συμφωνία με το Συμβούλιο έτσι ώστε οι ιδρυτικοί κανονισμοί τους να ανανεωθούν, να ενημερωθούν και να ευθυγραμμιστούν με την κοινή προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, European Labor Authority, είναι το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη και θα σας παρουσιάσω την πρότασή μου, δεν θα πω τώρα τίποτα. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης ε, και ζητάτε μια ευρωπαϊκή κάρτα ε, ε, ασφάλισης. Μέχρι τώρα δεν έχουμε προχωρήσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα κάνουμε σωστά αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα του νέου αριθμού ε, ευρωπαϊκού Κοινωνικής Ασφάλισης. Χρειάζεται όμως να διερευνηθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία, όλες οι λύσεις και να εκτιμηθεί το κόστος και η ωφέλεια. Ε, θέλει πολύ προπαρασκευαστική δουλειά αυτό. Ε, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θέλω να επαναλάβω ότι ήδη έχουμε πετύχει πολλά από κοινού. Ε, υπολογίζω στη δική σας δέσμευση και προσήλωση για να κλείσουν όλοι οι φάκελοι που ακρεμούν ακόμα μέχρι το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου σας και της Επιτροπής μας. Θα πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες μας, στις εκλογικές μας περιφέρειες, ότι είναι πραγματικότητα η κοινωνική Ευρώπη και για εκείνους. Περιμένω τώρα να συζητήσουμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Σας διαβεβαιώ ότι όλα τα μέλη της παρούσης Επιτροπής εργάζονται σκληρά. Έτσι, θα προωθήσουμε τα περισσότερα θέματα όσα περισσότερα μπορούμε. Τούτου λεχθέντος. Δίνω το λόγο στους συντονιστές. Ο κ. Ντέιβιτ Κάζα πρώτα από το ΕΛΚ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Κυρίως στον Επίτροπο τον κ. Ντομπρόφσκης και στην κυρία Μαρία Τάισεν που ήρθαν σήμερα το πρωί για την ανταλλαγή απόψεων αυτή αποτελεί τμήμα του διαθρωμένου διαλόγου. Πολλοί από εσά ίσως αναμένετε να πω κάτι για το θέμα της οροπίας ε, εργασίας και ιδιωτικής ζωής. Ακόμα συμβιβαζόμαστε όμως τις συμβαστικές τροπολογίες πάνω σε αυτό, οπότε καλύτερα να μην διακινδυνεύσω κάτι τις επόμενες ημέρες ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία επί των δυσχερεστέρων τομέων. Να πω όμως ότι το Κοινοβούλιο είναι στο πλευρό σας, κυρία Επίτροπε. Ενδεχόμενο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με το Συμβούλιο. Άρα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή. Η ερώτησή μου τώρα για την ε, κινητικότητα, την νομική κινητικότητα, το ελεκτικό συνέδριο, αρχές του έτους υπέβαλε έκθεση για την κινητικότητα των εργαζομένων, του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει των συστάσεων αυτών, να δραστηριοποιηθούν οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για φυστάμενα εργαλεία που αφορούν την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. Θα υπάρχει συνεργασία με τα κράτη-μέλη για τη βελτίωση συλλογή και χρήσεω δεδομένων για τι ροέ βάσει τη εργατική κινητικότητα. Και απασχόληση, αγορά εργασία ισορροπία και πώ η χρηματοδότηση η ευρωπαϊκή θα χρησιμοποιηθεί για την εργατική κινητικότητα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κάζα. Ο από, τη, από τους σοσιαστές. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι ήρθα σε αυτή τη συνεδρία της για να ακούσω την ισορροπία εργασία και ιδιωτική ζωή. Αλλά θα ήταν αγένεια κάτι τέτοιο για του φιλοξενούμενου μα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Εγώ είμαι περίεργη το θέμα αυτό τη οροπία εργασίας και ιδιωτική ζωής, αλλά σε άλλο βήμα θα συζητηθεί. Δύο ερωτήσει έχω. Κάποια στοιχεία αναφέρθηκαν, κάποια άλλα όχι. Σε ένα χρόνο περίπου έχουμε εκλογέ. Έχουμε πίεση χρονική να πετύχουμε πράγματα κυρίως στον τομέα της Επιτροπής μας. Κυρία Τάισον, έχω ερώτηση. Με τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, τι γίνεται. Από ό,τι άκουσα, είπατε ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Σωστή. Άρα συνεχίζεται η προετοιμασία. Τι εγγυήσει όμως έχουμε από εσά, τι εγγύσεις μας δίνετε ότι πράγματι θα υποβληθεί η πρότασή σας κατά διάρκεια αυτής της και αυτό στα πλαίσια της ε, κινητικότητας, του πακέτου για τη δίκαιη κινητικότητα. Δυστυχώς δεν υπήρχε τέτοια πτυχή το Μάρτιο. Τι εγγύηση μπορούμε να λάβουμε τώρα από σας για το πότε θα υποβληθεί πρώτα στο Κοινοβουλίο. Άλλη ερώτηση. Κάτι που δεν αναφέρατε αφορά η ερώτησή μου. Το, την εγγύηση για τα παιδιά θα θυμόσαστε ότι από την πρώτη μας ακρόαση με τη Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι σοσιαλιστές πίεζαν για μία εγγύηση για τα παιδιά. Έγινε, υπήρξε προπαρασκευαστική δράση για αυτή την εγγύηση για τα παιδιά. Θέλουμε όμως να αποκτήσει σάρκα και οστά σε αυτή την θητεία. Ερώτηση. Πότε θα εφαρμόσουμε τα μαθήματα που αντλήσαμε από την προπαρασκευαστική δράση όσον αφορά την εγγύηση για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουίκε Τρεμπέσιους που εκπροσωπεί το ECR έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπη, κύριε Ντομπρόφσης, κυρία Τάισεν. Στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία έχουμε κάποιες φιλόδοξες προτάσεις λάβει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορισμένες από αυτές βασίζονται και στη δήλωση προθέσεων για τα κοινωνικά δικαιώματα. Εν προκειμένου δύο ερωτήσει. Πρώτο, μιλούμε για τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Μέγα και φιλόδοξο έργο με σημαντικές δυσκολίες. Η σωστή νομοθεσία πρέπει να αποδείχνει την αξία της και στην καθημερινή πράξη, να μην επιβαρύνει πολύ τους εργαζόμενους και τους επιχειρηματίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα που πλησιάζει στο τέλος της κοινοβουλευτική περίοδος να αναλαμβάνεται τόσες πολλές νέες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες. Είδαμε ότι απέτυχε η κάρτα προσφορά υπηρεσιών. Δεν θα ήταν καλύτερα οι πρωτοβουλίε αυτέ να αρχίζουν νωρίτερα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο χρόνο για διαβουλεύσει και για εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Με τι καλύτερε των προθέσεων θα αποδειχθεί είτε επικίνδυνο είτε και λάθος να προσπαθήσετε δε και καλά να βγάλετε κάποια αποτελέσματα. Δεύτερη ερώτηση. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων οδήγησε σε πολλές νομοθετικές προτάσεις τις οποίες επεξεργαζόμαστε τώρα όπως η αρχή εργασίας, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ή πρόταση οδηγίας για διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων Ωστόσο είναι απλή δήλωση προθέσεων. Κάπου έχω την εντύπωση ότι πάτε να ξεφύγετε από το καθεστώς αυτό της δήλωσης προθέσεων και να περάσετε στους πολίτες ότι δήθεν αυτή η δήλωση προθέσεων είναι και καλά σοβαρή νομοθετική βάση. Δεν νομίζετε ότι ο κοινωνικός πυλώνας απέναντι στους πολίτες σε ό,τι αφορά δικαιώματα και υποχρεώσεις γίνεται λάθος αντικείμενο επικοινωνίας. Ευχαριστώ και αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω δύο άλλα πρόσωπα με δυσπρόφερτα ονόματα. Πηγαίνω αμέσως στην Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω την γλώσσα μου δανέζικα. Είμαι εδώ. Ευχαριστώ για τις εισαγωγικές σας τοποθετήσεις, θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο δεν θίξατε, ελπίζω να σχολιάσετε, δηλαδή του κοινωνικού πρωτοκόλου. Η ιδέα του κοινωνικού πρωτοκόλου είναι τα δικαιώματα των εργαζόμενων να εξισώνονται με την ενιαία αγορά και την ελεύθερη κυκλοφορία. Όλο και περισσότερες χώρες τα ζητούν αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη από το Γενάρη αποφάσισε ότι θέλουμε κοινωνικό πρωτόκολλο. Ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να αναμένουμε πρόταση για το κοινωνικό πρωτόκολλο. Μπορούμε να αναμένουμε πρωτοβουλία. Δεύτερη ερώτηση. Ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Έχετε κάποιο σχετικό χρονοδιάγραμμα. Μπορείτε να μας πείτε περίπου πότε θα κατατεθεί η σχετική πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ των Πρασίνων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε πρώτα. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτά που είπατε για τις καρκινογόνες ουσίες και τα καυσαέρια ντίζελ που έχουν βαριές συνέπειες σε ορισμένους τομείς της αγοράς εργασίας και βέβαια και στην υγεία του κοινού, στη δημόσια υγεία γενικότερα και πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Θέλω να θέσω ένα θέμα Ιδίω σχετικά με τον προπολογισμό και το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδίω τον κανονισμό Common Provision Regulation. Θέλω να πω ότι ορισμένες από τις οριζόντιες αρχές φαίνεται να αποδυναμώνονται. Αναμένω λοιπόν τα σχόλιά σας και τη δέσμευσή σας στο ότι θα διατηρήσετε τις αρχές της ε, εταιρικής σχέσης και της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ισότητας και μη διάκρισης. Η κυρία Τάισεν είπε ήδη μερικά θέματα σχετικά με την ισότητα φύλων. Προώθηση λοιπόν των αρχών ίσης μεταχείρισης φύλων, που βρίσκονται είναι πάρα πολύ σημαντικά εν προκειμένου, και βέβαιως και αηφόρο ανάπτυξη. Εξετάζουμε δηλαδή με ποιον τρόπο θα πρέπει να τα μεταφέρουμε αυτά στο μέλλον. Σχόλια επίσης παρακαλώ να κάνετε για το εάν θα κατατεθούν ισχυρότερες προτάσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με την συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα πρόσωπα με αναπηρίες όσον αφορά τις δαπάνες στο κοινωνικό τομέα του νέου πι. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω εκπρόσωπο της ομάδας EFDD, ούτε του ENF. Να δώσω το λόγο στους επιτρόπους και μετά έχω και άλλο μακρό κατάλογο προσώπων που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις. Αλλά ας δώσουμε πρώτα μια ευκαιρία να απαντήσουν στις πρώτες και μετά να συνεχίσουμε με τις επόμενες. Κύριε Ντομπρόσκης. Αξιότιμα μέλη, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα καλύψω κάποιες οριζόντιες ερωτήσεις και μετά η Μαριάν θα αναφερθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα πολιτικής και σχετικές προτάσεις. Η συνέχεια που θα δοθεί όσον αφορά την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, προβαίνουμε σε αξιολόγηση της σχετικής δράσης που βασίζεται στις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου κατά τη διάρκεια της περίοδου η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είχε προτεραιότητα στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό κρύβεται και πίσω από την πρότασή μας στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Εργατικού Δυναμικού που απασχολείται κυρίως με δυσυνοριακά θέματα. Σε κάποιο βαθμό καλύπτει τις εργασίες μας για την απόσπαση των εργαζομένων και άλλες πρωτοβουλίες. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού αντιμετωπίζεται. Θέλουμε δίκαιη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού είναι κάτι το οποίο είναι στο στόχαστο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθεί να είναι. Μετά τα ερωτήματά σας σχετικά με τον κοινωνικό πυλώνα, τις αρχές του πυλώνα αυτού, του κοινωνικού, και πώς θα ακολουθήσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αυτό ήταν το πνεύμα στο οποίο κινηθήκαμε. Και έτσι ανακοινώθηκε. Όταν διακηρύχθηκε στο Γκέτεμπορκ ο κοινωνικός ε, πυλώνας, υπήρξαμε σαφέστατοι. Ο κοινωνικός πυλώνας αυτός καθεαυτός εμπεριέχει διακηρύξεις αρχών. Δεν αναφέρεται σε δικαιώματα ή αξιώσεις θα δοθεί συνέχεια μετά από τις αρχές θα ακολουθήσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες είχαμε πει για την κοινωνική προστασία για όλους για δίκες συνθήκες εργασίας αυτές οι πρωτοβουλίες βασίζονται στις αρχές του κοινωνικού πυλώνα δεν βλέπω να υπάρχουν αντιφάσεις όσον αφορά τον αριθμό των νομοθετικών προτάσεων που έχουν προωθηθεί ή έχουν δρομολογηθεί να παρουσιαστούν πριν το τέλος της θητείας εσωτερικά όταν το συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό καθίσταται σαφές ότι η εντατικότητα υποβολής νομοθετικών προτάσεων θα μειωθεί πολύ σημαντικά μετά το Μάιο. Το Μάιο λοιπόν πρέπει να υποβάλουμε τις περισσότερες προτάσεις που ελπίζουμε να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ε, θητείας αυτής. Αναφερθήκατε επανειλημμένα ότι πλησιάζει το τέλος της θητείας. Πράγματι, από την άλλη πλευρά έχουμε ακόμα ένα χρόνο μπροστά μας. Και ένας χρόνος είναι μεγάλο χρονικό διάστημα αν εργαστεί κανείς εντατικά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα τους επόμενους μήνες να επικεντρωθούμε λιγότερο επί νέων πρωτοβουλειών και περισσότερο επί ολοκληρώσεως δρομολογηθήσεων πρωτοβουλειών. Σχετικά με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον κανονισμό κοινές διατάξεις συνεχίζεται το έργο. Δεν λέω ότι θα αποδυναμωθούν οι φυστάμενες οριζόντιες αρχές εμπεριέχονται ένα στοιχείο όπως η ενίσχυση της σχέσης με τις διαθετικέ μεταρρυθμίσεις, με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και συμπερίληψη αυτών των πτυχών και απλούστευση ενδεχομένω των διοικητικών απαιτήσεων, ούτω ώστε αυτά τα προγράμματα να μπορούν να εφαρμοστούν πιο εύκολα, για να διευκολύνει την πρόσβαση. Ελπίζουμε η τελική πρόταση να είναι ισορροπημένη συγκεκριμένη ερώτηση που ετέθη για τα καρκινογόνα και τα καυσαέρια από διζελοκινητήρες. Θέλουμε να επικαιροποιήσουμε την οδηγία για μεταλλαξιογόνα και καρκινογόνα ε, ε, και αφορά τα χημικά, τις χημικές ουσίες στον τόπο εργασίας και έχουμε σχετικές προτάσεις που θα βασίζονται επί εξελισσομένων επιστημονικών στοιχείων. Μέχρι τώρα δεν είχαμε αρκετά στοιχεία και πληροφορίες για να συμπεριληφθούν οι εξατμίσεις από τις ζελοκινητήρες. Συνεχίζονται οι μελέτες για να περιστεί έκθεση στις εξατμίσεις ε, από τις ζελοκινητήρες στο χώρο εργασίας. Ευχαριστώ. Ε, Κυρία Τέσσερα, ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Για την κινητικότητα των εργαζομένων, να τα πω ολλανδικά καλύτερα. Βεβαίως, έχουμε και διερμηνία. Περισσότερα από πουθενά. Να την αξιοποιήσω. Σας ευχαριστώ για την ευελιξία σας. Λοιπόν, η κινητικότητα των εργαζομένων και η ΕΛΑ, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας πραγματικά λάβαμε υπόψη τις ε, παρατηρήσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Δημοσιεύθηκε η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου πριν κάνουμε εμεί τη δική μας πρόταση για την Ευρωπαϊκή Αρχή τη πριν τη λανσάρουμε και την παρουσιάσουμε. Και πραγματικά ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη οι παρατηρήσεις τους ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πύλη Γιούρε και ε, ε, άλλα σχετικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα. Και να συνειδητοποιήσουν καλύτερα οι άνθρωποι ποιε είναι οι δυνατότητέ του και τα δικαιώματά του στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Πραγματικά, σε ό,τι αφορά τον αριθμό κοινωνική ασφάλιση. Χρειάζεται περισσότερο χρόνο από ό,τι είχα φανταστεί και εγώ ίδια ότι θα χρειαζόταν όταν θα το παρουσιάσουμε θα πρέπει να είναι ένα σωστό, καλά προετοιμασμένο σχέδιο με τεχνική πληροφόρηση. Θα πρέπει να συλλέξουμε τώρα ακόμα αυτές τις τεχνικές πληροφορίες για να δούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατότητα και να είναι και αποτελεσματική. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε με νομοθετική πρόταση ή με άλλες μεθόδους. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει καν στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουμε και θα λανσάρουμε πανευρωπαϊκά αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση με συγκεκριμένη πρόταση. Τι πρόταση θα είναι αυτή δεν ξέρουμε ακόμα, όποια και να είναι επικοιτακόμαστε, είμαστε στη διερεύνηση για τον αριθμό κοινωνική ασφάλιση. Μην λέτε ότι έχει εγκαταληφθεί καθόλου, είναι επιτάπητο. Απλώ το μελετούμε και προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια τη ηττία αυτή, αλλά κυρίω όταν φέρουμε την πρόταση να είναι πρόταση κανονική, ε, καλά προετοιμασμένη, που να μπορεί να πατήσει τα πόδια τη και να μπορέσουμε και ηλεκτρονικά να τα εφαρμόσουμε στην ψηφιακή εποχή. για τις καρκινογόνες ουσίες και τον ντίζελ. Συνεχίζονται οι διάλογοι τριμερείς και οι συνομιλίες. Το ντίζελ δεν έχει συμπεριληφθεί ακόμα γιατί δεν είχαμε τα επιστημονικά δεδομένα και η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν είχε καταλήξει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ουσιών. Ωστόσο, στο μεταξύ, σε διάφορα κράτη-μέλη λαμβάνονται αποφάσεις μεταξύ αυτών στην Γερμανία και στην Αυστρία. Γίνονται και με επιστημονικές έρευνες και μελέτες και έχουν έρθει αυτά και στον τριμερή διάλογο. Αν καταφέρει το Κοινοβούλιο να πείσει το Συμβούλιο, σίγουρα εμεί θα παίξουμε ένα ρόλο υποστηρικτικό. Είμαστε πάρα πολύ θετικοί σε αυτή την πρόταση και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια λύση στον τρέχοντα τριμερή διάλογο. Αυτό είναι θέμα των δύο συνομοθετών. Εμείς πάντως θέλουμε ε, να συμπεριληφθεί. Έχουμε νέα επιστημονικά δεδομένα. Αν θα φέρουμε νέες προτάσεις, ρωτήσατε. Με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για πρόσωπα με αναπηρία. Όχι ακόμα νομοθετική πρόταση δεν πρόκειται ε, να φέρουμε καινούρια που να μην έχει εξαγγελθεί και που να μην είναι στο πρόγραμμα εργασιών μας. Ωστόσο, εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά στην νομοθετική πρόταση για την προσβασιμότητα, που και αυτό είναι ε, σχετικό με τη σύμβαση του ΟΗΕ για τα ατομαμένα πυρίες. Αυτό θέλουμε οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί γιατί θα βελτιώσει πολύ τη ζωή των 80 εκατομμύριων ανθρώπων που έχουν αναπηρίες. Και στο μέλλον θα είναι ακόμα περισσότεροι γιατί γυράσκει ο πληθυσμός. Σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων και τη βυσμή διακρίση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε υπόψη σε όλες τις προτάσεις μας. Ε, αφορά θεμελιώδη βασικά δικαιώματα έχουμε και δευτερογενή ε, βέβαια νομοθεσία και θα πρέπει να φροντίζουμε να γίνονται σεβαστοί οι κανόνες και να τηρούνται. Και μας ενδιαφέρει και το παρακολουθούμε. Τι άλλο θα κάνουμε, λέτε, στο επόμενο διάστημα όσο απομένει. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης. Έχουμε ένα χρόνο ολόκληρο ακόμα. Ε, επίσης υπάρχουν και προγράμματα εργασίας ε, για το διάστημα αυτό λέμε big on the big things και small on the small things, δηλαδή να είμαστε ε, σε θέση να αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που πρέπει τα προβλήματα, ε, τα μεγάλα και τα σπουδαία με μεγάλη προσοχή και λιγότερο τα μικρά. Είναι πολύ διάστημα ένας χρόνος, πολύ μεγάλο. Και εγώ έχω μάθει στο κοινοβούλιο εδώ ότι δουλεύουμε μέχρι την τελευταία μέρα. Οπότε έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις ε, σωστά. Τι άλλο. Την εγγύηση για τα παιδιά. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας υπηρεσιακό. Στις 16 Απριλίου δόθηκε αυτό. Με κατευθυντήριες γραμμές και δράσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δείτε, δεν ξέρω μήπως δεν είχατε χρόνο να το κοιτάξετε, ε, αλλά στη λίστα με τις συστάσεις αναχώρα που εκδόθηκε χθες, Εχθές μάλιστα αποφασίστηκε κιόλας και δημοσιεύτηκε. Ε, κάνουμε συστάσεις για το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά ε, και τη φύλαξη των παιδιών. Στο παρελθόν αυτό δεν ήταν κάτι που είχε γνώρισει μεγάλη προσοχή. Και επιτρέψουμε να σας θυμίσω κιόλας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πιλωτικό πρόγραμμα, πιλωτική δράση ακριβώς βάσει της πρότασης του Κοινοβουλίου για την εγγύηση για τα παιδιά. Νομίζω απάντησα εδώ σε σημαντικότερα ερωτήματα και σταματώ, Πρόεδρε. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Θα παραμείνετε, κυρία Τάισεν. Ο κύριος Ντομπρόφσκης είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει. Ευχαριστώ που απάντησε τουλάχιστον στο πρώτο μέρος των ερωτήσεων. Ίσως μπορούμε να σας υποβάλουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά είπατε ότι σας ενδιαφέρει η υλοποίηση των υπεσχημένων. Αναμένουμε λοιπόν την υλοποίηση. Τώρα, θα δώσω το λόγο στους υπολείπους ε, βουλευτές που ζήτησαν το λόγο. Κύριε Πυρίνσκι, είστε πρώτος στον κατάλογο μου τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βέβαια την ερώτησή μου ήθελα να την κάνω στον Αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόφσκης. Δεν θέλω όμως να διακόψω την ορμή με την οποία αποχωρεί τις αιθούσεις. Θα εμπιστευτώ λοιπόν την Επίτροπο κυρία Τάισιν να τον ευαισθητοποιήσει γιατί εγώ θα στείλω γραπτό στην ερώτηση αφού νομίζω ότι άπτεται των δικών του αρμοδιοτήτων και έχει σχέση με τον κοινωνικό διάλογο, την κοινωνική εταιρική σχέση και τις συλλογικέ συμβάσεις. Κυρία Πρόεδρε, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και η ίδια η Επίτροπος τόνισαν τη σημασία της προώθησης της κοινωνικής Ευρώπης σε όλες τις πτυχές της. Και τα δικαιώματα που περιέχονται στον κοινωνικό πυλώνα. Εγώ θέλω να έρθω στα δικαιώματα υπαριθμών 6 και 8. Το 6 αναφέρεται στις αμοιβέ. Λέει ότι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε δίκαιες αμοιβέ που να επιτρέπουν αξιοπρεπή διαβίωση και ότι αυτές θα ρυθμίζονται με τρόπο προβλέψιμο σύμφωνα με τις ε, εθνικές πρακτικές και τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων. Το 8 λέει ότι οι κοινωνικοί εταίροι ενθαρρύνονται να διαπραγματεύονται και να συνάπτουν συλλογικέ συμβάσεις για θέματα που τους αφορούν με σεβασμό βέβαια της αυτονομίας τους. Όλα αυτά περιέχονται και στην αιτιολογική σκέψη 20 που λέει πολύ καθαρά ότι ο κοινωνικός διάλογος παίζει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού και ότι οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν σημαντικό ρόλο για ε, την εφαρμογή των προβλέψεων του πυλώνα με την διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων και με τις συλλογικές δράσεις. Στην διάρκεια της προετοιμασίας μας για τον ε, διαθρωμένο διάλογο είχε υπάρξει και ένα θέμα στο τέλος της λίστας των προτάσεων από ορισμένου συναδέλφου μα που ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει τη λιτότητα και να ξαναχτίσει το σύστημα συλλογικών συμβάσεων. Η ερώτησή μου προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής θα ήταν βλέπει την ανάγκη να επανικοδομηθεί το σύστημα συλλογικών συμβάσεων διότι γνωρίζουμε όλοι ότι από την κρίση του 2008 έχει διαβρωθεί το σύστημα των συλλογικών διαπραγματεύσεων με σοβαρές επιπτώσεις μείωσης της ε, δικαιοσύνης στις ρυθμίσεις για τις, δηλαδή του δίκαιου χαρακτήρα δηλαδή των αμοιβών και αυτές οι συνέπειες τελικώς οδήγησαν σε αύξηση των ανισοτήτων που αποτελεί σημαντική πρόκληση νομίζω και για το μέλλον των πόλης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για να μην μακρηγορώ. Πιστεύω ότι ο αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης στο χαρτοφυλάκιο του οποίου μπαίνει και η σχέση των κοινωνικών εταίρων παρέλειψε να εξηγήσει στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή πώς βλέπει την διαδικασία ώστε να υλοποιηθούν τα δίκαια που προβλέπει ο κοινωνικό πυλώνα. Μίλησε για την ανάγκη νομοθεσία ώστε τα δικαιώματα να μεταφερθούν στην πραγματικότητα. Όμω, στο κεφάλαιο 14, το οποίο διαπραγματευθήκαμε με το Συμβούλιο, λέει ότι για να είναι νομικά εξαναγκαστά τα δικαιώματα αυτά, Χρειάζονται πρώτα συγκεκριμένα μέτρα και νομοθεσία. Μέτρα λέει. Και τα μέτρα βέβαια είναι προνόμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών μελών. Όμως σίγουρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίζει το ρόλο του μοχλού για την προώθηση της εφαρμογής των προβλέψεων του πυλώνα. Όπως είπα λοιπόν, αυτά θα τα βάλω όλα σε μια γραπτή ερώτηση που θα διαβιβάσω στον Αντιπρόεδρο. Όταν μιλεί όμω για σύγκριση προς τα πάνω, για ευρωπαϊκό εξάμεινο κλπ, χωρίς να αναφέρει τον κοινωνικό διάλογο και τις συλλογικέ συμβάσει. θεωρώ ότι είναι σημαντική παράληψη στην προσέγγιση του Αντιπρόεδρου των και επομένω της Ευρωπαϊκή Επιτροπής στο σύνολό τη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, αλλά σε ό,τι αφορά τώρα το πι στην περίπτωση όπου το ESF συν είναι απολύτως συν, αυτό μάλλον είναι σημαντικό ερώτημα. Οι δε προτάσεις μας για τον διαθρωμένο διάλογο θα αναφερθούν στην ανάγκη να διατηρηθούν οι λειτουργίες των διαφόρων ταμείων με προσαρμογές αλλά να μην χαθούν οι βασικές λειτουργίες υπέρ αυτών που βρίσκονται σε βαριές συνθήκες φτώχειας και να τα χώσουμε όλα αυτά τώρα σε ένα ενιαίο ταμείο απειλεί νομίζω τη λειτουργία αυτών των δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Έχω το αίσθημα ότι, την αίσθηση μάλλον, ότι αυτό το θέμα είναι μάλλον δική σας αρμοδιότητα κυρία Τάισιν. Ίσως μπορείτε να κάνετε μια προσπάθεια να απαντήσετε, μιας και ο κύριος Τομπρόφσκης απεχώρησε. Γιατί τα θέματα αυτά ε, είναι, ε, σας είναι πολύ γνωστά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας δώσω μια πρώτη απάντηση, θα προσπαθήσω, αλλά φυσικά ρωτήστε γραπτό στον Αντιπρόεδρο, θα τον ενημέρωσουμε κι εμείς. Σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς εταίρους, πρέπει να σας πω ότι τούτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι οι επίτροποι λαμβάνουν πολύ σοβαρά το ρόλο τους. Και όλα αυτά δεν είναι θεωρίες, είναι ε, πολιτική, κανονική. Τι κάναμε στην αρχή, το πρώτο έτος της θητείας μας ε, παρουσιάσαμε μια νέα προσέγγιση για τον κοινωνικό διάλογο γιατί είδαμε ότι μετά την κρίση ο κοινωνικός διάλογος δεν ήταν πώς να το πω, τόσο ανθυρός σε όλα τα κράτη-μέλη παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμφωνήσαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει και αυτό εφαρμόζουμε. Δράσεις λοιπόν αυτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αιτήματα στα κράτη-μέλη αλλά και ε, ενδυνάμωση και χειραφέτηση των κοινωνικών εταίρων. Τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε τριμερείς κοινωνικές συνόδους ε, κορυφής. Εγώ είμαι πάντα εκεί παρούσα και η κυρία Ολσκοκ ε, από πλευράς Κοινοβουλίου και πραγματικά έχει γίνει αλλαγή ουσιαστική ε, γίνεται διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και δεν είναι μια ευγενική αλληλογραφία ε, τυπική. Γίνονται πολύ σοβαρές συζητήσεις με κοινή ατζέντα όλοι παρόντες. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει ο μακροοικονομικός διάλογος επίσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Υποσχεθήκαμε και το υλοποιούμε από κοινού και δεν διαμαρτύρονται οι κοινωνικοί εταίροι γι' αυτό. Δεν παραπονούνται. Ε, τους διαβουλευόμαστε για μεγάλα πολιτικά ζητήματα, είτε είναι η ενέργεια αυτό, είτε κάποια άλλα, γιατί έχει αυτό επιπτώσεις φυσικά ακόμα και ε, στον τόπο εργασίας και γενικότερα φορά πολλούς εργαζομένους και εκείνοι εκπροσωπούν πολλούς. Και βέβαια για τα κοινωνικά θέματα πάντα έχουμε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. εξασφαλίσαμε πολύ καλύτερη συμμετοχή τους ε, στην άσκηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τους ενημερώνουμε και γίνεται διαβούλευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν ε, εκδοθεί η ετήσια μελέτη για την ε, γέννηση της οικονομίας έχουμε τακτικές επαφές και συναντήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους και πριν προβούμε στις εκθέσεις, στην έκδοση των εκθέσεων αναχώρα διαβουλευόμαστε με τους κοινωνικούς εταίρους επιτόπου στην κάθε χώρα μέλος. Είτε η ίδια επίτροπη είτε κάποιοι υπάλληλοι για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που έχουμε σε όλες τις χώρες πλέον στις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, ζητούμε από τις χώρες στην έκθεση αναχώρα και στις συστάσεις αναχώρα να ενθαρρύνουν τον κοινωνικό διάλογο και να τον ακούν και να εισακούν. Ξέρω και τα ξέρω απ' έξω ότι υπάρχουν δύο κράτη-μέλη όπου έχουμε πολύ συγκεκριμένη αναφορά, όχι σε ιδεολογικές σκέψεις και τα λοιπά, στις συστάσεις αναχώρα. Σύσταση να συνεργάζεστε καλύτερα με τους κοινωνικούς εταίρους και καλύτερο θεσμικό πλαίσιο να δημιουργήσετε και περισσότερο χρόνο για τη διαβούλευση. Σε εθνικό επίπεδο σας τα είπα, ότι παρακολουθούμε κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης πώς γίνεται αυτό, τη δημιουργία ικανοτήτων και υποστηρίζουμε αυτό το capacity building των κοινωνικών εταίρων και στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα υπάρχει και αντίστοιχη χρηματοδότηση με τις υπηρεσίες, τις υποστηριστικές και το αντιπρόεδρο που αναφέρατε. πραγματικά μας απασχολεί πάρα πολύ σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουμε δηλώσει από την αρχή και υλοποιούμε τις προτάσεις αυτές. Εκπλήσωμαι λίγο που ακούω τέτοια σχόλια. Γιατί δεν καταλαβαίνω σε τι αναφέρεστε. Εγώ τα αντίθετα βλέπω. Βεβαίω πάντα χωράει βελτίωση και στα κράτη-μέλη και παντού γιατί τους το ζητάμε άλλωστε. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το υποστηρίζει και θα λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία του κοινωνικού πυλώνα. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, ESF+. Την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε τη συγκεκριμένη πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού. Ναι, θέλουμε ένα ESF+, τώρα. Και ομολογώ εγώ την ενοχή μου, γιατί εγώ τους πίεσα να το κάνουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να επενδύσουμε καλύτερα στους ανθρώπους, στο ανθρώπινο κεφάλαιο ε, με την ευρύτερη έννοια. αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε χρήματα για εκείνους που θα χρειάζονται περισσότερο. Θα έρθουν οι προτάσεις την επόμενη εβδομάδα και με το καλό θα τα συζητήσουμε. Δεν είναι όμνιμπους να κάνουμε ό,τι θέλουμε τα λεφτά του κοινωνικού ταμείου. Αγωνιστήκαμε γι' αυτά. Έχει μεγαλύτερο μερίδιο τώρα ε, στην συνοχή από ό,τι στο παρελθόν γιατί το χρειαστήκαμε δεν είχαμε μόνο προβλήματα σύγκληση στην Ευρώπη που υπάρχουν και παραμένουν και χρειάζεται δουλειά εκεί και με λεφτά από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, αλλά θα πρέπει να επενδύσουμε στι δεξιότητε και αυτό είναι πρόβλημα παντού στην Ευρώπη. Και θα φροντίσουμε να πιάσουν ε, όσο γίνεται περισσότερο τόπο τα χρήματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Σωσοπάβελ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ για το χρόνο σας, για τις απαντήσεις σας. Ερωτήσεις. Έχω δύο-τρεις ερωτήσεις. Αφορούν κάποια θέματα. Καταρχάς, ο συντονισμός του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ε, τελεί υπό διαπραγμάτευση. Αλλά ανησυχώ. Μήπως εθνικό δίκαιο λάβουν μέτρα τα κράτη-μέλη το θέμα αυτό των επιδομάτων της οικογένειας. Μία από αυτές είναι η Αυστρία ε, που θα αναλάβει 1η Ιουλίου την Προεδρία του Συμβουλίου όταν μιλάμε για ίσες αμοιβέ για ίδια εργασία, πρέπει να είμαι και για ίδια ευεργετήματα για την ίδια εργασία στον ίδιο τόπο. Ποια είναι η απόψη από αυτού, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά των μέτρων που αναφέρονται στην εθνική νομοθεσία κάποιων κρατών που κάνουν διακρίσεις όσον αφορά τους εργαζομένους, κατά την άποψή μου. Δεύτερο, να τονίσω και αυτό που είπε η κεφαλής της ομάδας, η Άγνες, για τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρατε. Είναι σημαντικότατο να διευθετηθεί το θέμα σε αυτή τη θητεία. Δεν μπορούμε να περιμένουμε, αποτελεί προτεραιότητα. Πρέπει να λυθούν κάποια προβλήματα. Έχω πλήρη επίγνωση αυτού. Πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Πρέπει να βρούμε σωστή λύση και το ταχύτερο δυνατόν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει σε αυτή τη θητεία και να εφαρμοστεί το μέτρο πλήρω το ταχύτερο τη δυνατόν, διότι μπορεί να επιλύσει σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει στην Ευρώπη. Τέλο, κάτι εξίσου σημαντικό, έχω δέκα δευτερόλεπτα. Είμαι απογοητευμένο. Γιατί διπλασιάστηκε μόνο το έρασμο συν. Εγώ θα πολεμούσα για τουλάχιστον τριπλασιασμό του ποσού. Κάτι που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Και ελπίζαμε ότι και εσεί θα υποστηρίζατε αυτό το μέτρο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο λεπτά έτσι δεν είναι. Ο συνάδελφος Σπυρίνσκι, τον οποίο εκτιμώ πολύ νομίζω κάπως το παράκανε. Έξι λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Εγώ θα κρατήσω τα δύο λεπτά. Ήθελα να μιλήσω για την οδηγία για την απόσπαση εργαζόμενων. Αρχές της εβδομάδας μάθαμε ότι το θέμα δεν θα συζητηθεί τον Ιούνιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ήδη τον Μάιο, δηλαδή στην επόμενη περίοδο συνόδου, τη επόμενη εβδομάδα. Στην Επιτροπή Απασχόλησης είχα, είχαμε 38 ναι και 14 όχι, δηλαδή ήταν και τεράστια η πλειοψηφία. Αλλά γενικά δεχόμαστε. Τώρα, υπάρχει το ζήτημα των ταξιδιών επαγγελματικών ταξιδιών, ταξιδιών υπηρεσίας, αποστολών υπηρεσίας. στη Γαλλία και στο Βέλγιο δυσχεραίνονται τα ταξίδια αυτά, διότι πρέπει κανείς να καταθέτει τα έγγραφα από πριν. Και αν δεν το κάνει, τότε πέφτουν κυρώσει. Αυτή η ρύθμιση υποτίθεται έχουν διατηρηθεί. Εμείς δεν το βρήκαμε όμως, δεν τα βρήκαμε, παρόλο που εξετάσαμε προσεκτικά. Η ρύθμιση των οκτώ ημερών εξακολουθεί να είναι ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθεί να είναι εγγυημένη ή όχι, διότι είναι σημαντικό. Έχω λάβει άφθονες επιστολές από μικρές και μεσές επιχειρήσεις που μου λένε ότι δεν είναι δυνατόν. Πρόκειται για απλές κανονικές αποστολές, δεν είναι, δηλαδή ταξίδια υπηρεσιακά, δεν είναι απόσπαση εργαζομένων. Χρειάζεται λοιπόν να το ξαναδούμε αυτό, ώστε να το αλλάξουμε στην αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων. Κάποια δευτερόλεπτα μου μένουν, έρασμος συν. Εδώ νομίζω πραγματικά πρέπει να υπάρξει κάποια κίνηση. Αγαπητή Μαριάν, έρασμος συν. Πρόκειται πραγματικά για το σήμα κατατεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάντε μια προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει ο κόσμος να αντιληφθεί ότι κάνει καλό η παραπάνω Ευρώπη και δεν είναι απαραίτητα καλή η λιγότερη Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Μάν. Ο κύριος Ζαϊρανόπουλος, έχει το λόγο. Ε, ας δούμε για ποια κοινωνική Ευρώπη μιλάμε. Με παράδειγμα την ε, Ελλάδα. Χθε το πρωί ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, πανηγύριζε στην Ελληνική Βουλή ότι τον Αύγουστο του 2018 η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια και απαλλάσσεται από την εποπτεία των θεσμών. Κυρία Τάισεν, είναι αλήθεια αυτό. Γιατί χθε το βράδυ ανακοινώθηκε η συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τους θεσμούς από την Κομισιόν, η οποία από ό,τι βλέπουμε προβλέπει νέα μέτρα, αντιλαϊκά βεβαίως, το 2019, 20, 21, 23, δηλαδή πολιετής δεσμεύσεις για πολύ μετά από το μνημόνιο και χωρίς χρονικό ορίζοντα. Όχι απλώς διατήρηση των μέτρων, αλλά και δέσμευση να ληφθούν νέα μέτρα χωρίς χρονικό ορίζοντα, αν αλλάξουν τα δεδομένα. Όπως επίσης και δέσμευση των ελληνικών, της ελληνικής κυβέρνησης ότι πριν πάρει οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία θα παίρνει την έγκριση των θεσμών. Δεύτερο, μιλάει για πλεονάσματα 3,5% δημοσιονομικά μέχρι το 2023 και 2,5% μέχρι το 2060. Αυτά από ό,τι καταλαβαίνετε βγαίνουν από τους φόρους. Όταν λοιπόν η φορολογία των επιχειρήσεων μειώνεται με συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Κυβέρνησης, ποιος αλήθεια θα πληρώσει αυτούς τους αυξημένους φόρους. Εδώ αναφέρομαι στο αφορολόγητο, που, τη μείωση του αφορολόγητου που χτυπάει τα φτωχότερα στρώματα και που φαίνεται ότι από το 2020 έχετε πιο μπροστά το 2019. Επίσης, ιδιωτικοποιήσεις, πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Και ρωτάω την κυρία Τάισεν, είναι και οι οργανισμοί ίδρευσης Αθήνας και Θεσσαλονίκης μέσα από το πρόγραμμα. Και τελευταίο, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ως γνωστόν με το μνημόνιο καταργήθηκαν στην Ελλάδα πλήρως μιλάνε για ε, αποκατάσταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, αλλά με έναν όρο, ότι θα επιτρέπεται από την υψηλή κερδοφορία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Αλλιώτικα δεν μιλάμε για αυξήσει. Αυτό είναι συλλογική σύμβαση. Και τέλο, ε, το ίδιο κείμενο τη Επιτροπή μιλάει για συνέχιση χωρί χρονικό ορίζοντα των περικοπών των συντάξεων που ήδη έχουν κοπεί πάνω από 17 φορέ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, για πολύ μετά από το, τέλος, το τυπικό τέλο του μνημονίου τον Αύγουστο του 2018. Ορισμένε απαντήσει με κέντρο αν τελικά θα σταματήσει η εποπτεία μετά το 2018 ή όχι. Thank you. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Εντουάρ Μαχτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εντουάρ με λένε, ναι, το μικρό. Κάνετε εξαγγελίε ένα χρόνο πριν το τέλο τη θητεία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιταχύνει για τον κοινωνικό ορίζοντα. Βέβαια δεν θα διαμαρτυρηθούμε. Στο μυαλό σας υπάρχουν και τακτικισμοί. Γιατί το ε, τριπλό α το κοινωνικό προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε, να το εξασφαλίσουμε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θέλουμε ποιοτικά κείμενα και όχι ποσοτικά. Προσοχή. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Εγώ δεν θέλω να καταδικάσω την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναφερθήκατε για την ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Θέλω να τονίσω εδώ την υποκρισία των κρατών μελών. 14 που κήρυξαν αντάρτικο για να μην περάσει αυτή η οδηγία και είμαι πάρα πολύ ε, θυμωμένος, έξαλλος για να μην πω τίποτα παραπάνω που η χώρα μου πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια. Ελπίζω να μην ενδώσετε και να φροντίσετε αυτή η, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών να περάσει. Και η, διάσταση του γονέα δεν είναι μόνο η μητέρα και ο πατέρας στην οικογένεια. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην μας αδειάσει. Τουλάχιστον εμείς δεν θα υποχωρήσουμε. Να πω και κάτι ακόμα που θέλω να επισήσω την προσοχή σας αυτό, η δίκαιη μετάβαση. Και μιλήσατε για το ρόλο των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των κοινωνικών εταίρων. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη μεταρρύθμιση του συστήματος ETS για την εμπορία εκπομπών δεν είναι δικό σας χαρτοφυλάκι, αλλά θελήσαμε να υπάρχει μια εποπτεία, μια διαχείριση σε τοπικό επίπεδο με τους κοινωνικούς εταίρους, ΟΤΑ κτλ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το θέλησε. και μιλάμε για ένα ταμείο για τη δίκαιη μετάβαση και εσείς μιλήσατε για τον εξυγχρονισμό. Μα ποια θέση θα έχουν εκεί οι κοινωνικοί εταίροι, τι δουλειά έχουν με τον εξυγχρονισμό. Πολύ ωραία ενεργειακή μετάβαση και συμφωνώ, αλλά δεν πρόκειται να πείσετε Πολωνούς ή άλλους ανθρακορίχους ότι κοιτάξτε θα κλείσουν τα ορυχεία και θα δούμε μήπως χτιστεί τίποτα δίπλα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της και πριν κλείσουν τα ορυχεία να δημιουργηθεί εναλλακτική δραστηριότητα. Επίσης, βλέπετε σήμερα τι γίνεται στην επικαιρότητα, στην κρίση με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Διαπραγματευόμαστε για μια διήθηση, ένα φιλτράρισμα των εξωτερικών ξένων επενδύσεων και έχω αγανακτήσει με τη θέση των ε, Υπουργών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ορισμένων συναδέλφων που δεν θέλουν να ακούσουν λέξη. Η Κίνα θα έρθει εδώ μαζικά να επενδύσει στις πολύ υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις και εμείς θα το χάσουμε το παιχνίδι. Και ο Τραμπ θα μας ε, απαγορεύσει να πουλάμε εκεί το χάλιβά μας και μετά θα χάσουμε και τον έλεγχο τους Κινέζους. Και τελειώνω. Κυρία Τάισεν, Κάπως με ενόχλησε αυτό που είπατε για την ε, ε, ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Είπατε ότι θέλετε όλοι να σέβονται τους κανόνες και σας παραθέτω. Τι θα πει επιθυμώ. Ε, ε, ε, απαιτώ. Εσείς είπατε επιθυμώ. Τι επιθυμείτε. Όταν πρόκειται για οικονομικέ κυρώσει, απαιτείται και τιμωρείται με κυρώσει. Όταν πρόκειται για την ισότητα ανδρών και γυναικών, είναι επιθυμία. Καθόλου επιθυμία. Απέτηση είναι η δικιά μου. Ευχαριστώ κύριε Μάρτα. Ο κύριος Μπαλάς. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε να συζητήσετε μαζί μας σήμερα. Δυστυχώς δεν άκουσα την αρχική παρέμβασή σας, παρουσία του Επιτρόπου Ντομόσκη. Ζητώ συγγνώμη, δυστυχώς καθυστέρησα λίγο. Δεν θα θέσω λοιπόν ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Έχω δύο θέματα να θέσω. Το πρώτο, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Προσωπικά σας υποστηρίζω είναι σημαντικό. Όπως οι σοσιαλιστές είπαν και όπως ο κ. Πάβελ ανέφερε προηγουμένως, υποστηρίζουμε την ιδέα μιας κάρτας κοινωνικής ασφάλισης ευρωπαϊκής, διότι πρέπει να έρθει ένα παράδοξο. Πολλοί από τους συναδέλφους, κράτη-μέλη, δεν θέλουν να κινητοκοπήσουν το θέμα και να έχουν ευρωπαϊκό επίπεδο κοινωνική ασφάλιση, λέγοντα ότι αυτό είναι ρόλο των κρατών μελών. Και όταν προσπαθούμε να κάνουμε συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση, είμαι συντονιστή για αυτήν την έκθεση, τι βλέπουμε. Ότι δεν κάνουν τη δουλειά του σαν κράτη-μέλη. Είτε όσον αφορά του ελέγχου, είτε αφορά τη διοικητική δυνατότητα, αδειοδότηση μετακινήσεως για την κινητικότητα των εργαζομένων. Οπότε ποια είναι η κατάσταση. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες οι οποίοι ε, κινούνται και δεν βρίσκουν διοικητικές απαντήσεις στο θέμα τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ισχυροποιηθούν κάποια εργαλεία ε, ελέγχου για την κοινωνική ασφάλιση για να υπάρχει ισοδυναμία μέσω της κινητικότητας των εργαζομένων, κάτι που έχουμε συμπεριλάβει στα μέτρα μας και απ' την άλλη με την ισότητα της αντιμετωπίσεως, με την κοινωνική προστασία των κινουμένων, μετακινουμένων εργαζομένων. Διότι με την παρούσα κατάσταση δύσκολα συνδέονται τα δύο. Και έχω μια ερώτηση. Πότε πραγματικά θα ψηφιοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την κινητικότητα των εργαζομένων όπως είναι η ESSE, η πλατφόρμα που ανακοινώσατε εσείς για το 2019. Δεν είναι κάτι απλώς με τεχνική. Είναι κάτι σημαντικό αν ψηφιοποιήσουμε τι διαδικασίε όπω γίνεται η ανταλλαγή πληροφοριών που υπάρχει στο Βέλγιο, ε, με το ε, τράπεζα ε, Καφούρ, με, το, με, το, με την βάση δεδομένων Μιμόζα κλπ. Θα επιταχύνουμε την κοινικότητα των εργαζομένων με καλύτερη προστασία ταυτόχρονα θα έχουν περισσότερε πληροφορίε και η έλεγχη θα είναι πολύ πιο εύκολοι. Σαν εισηγητή όσον αφορά τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφαλίσεω, χρειάζομαι αυτέ τι πληροφορίε σήμερα, ούτω ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να εργαστεί με έναν τρόπο σωστό όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν θα μακρηγορήσω κι άλλοι ερώτηση για τους συνοριακούς εργαζομένους, αλλά για το εσύ και τη διαδικασία των διαδικασιών που θα καταλήξει σε αριθμό και στους ασφαλίσεις κάποια μέρα, χρειαζόμαστε σήμερα εχέγγυα ε, διαβεβαιώσεις από την πλευρά σας, ε, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας. Ο κύριος Ντομπρόσκης και η κυρία Τάισαν είπαν ότι πράγματι ήρθε η ώρα για αποτελέσματα. Αυτό είπαν. στην αρχή της συζήτησης. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι περνάει ο χρόνος και δεν έχουμε τόσα μεγάλα χρονικά περιθώρια για λήψεις αποφάσεων. Πρέπει να υπάρξουν αποτελέσματα πριν τις επόμενες ευρωεκλογές. Τούτων λεχθέντων θα δώσω το λόγο σε εσά κυρία Τάισεν. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις όμως που ήταν σχετικές η μία με την άλλη. Προσπαθήστε παρακαλώ να απαντήσετε όσο δυνατόν περισσότερο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Και πάλι στα Ολλανδικά μου επιτρέπετε. Um, just a Λοιπόν, πρώτα ε, τα οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα τέκνων. Γνωρίζετε την άποψή μου, είναι πολύ σαφής ε, για το τι σημαίνει και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή πρόταση, ευρωπαϊκή βάση, δεν θέλουμε να ε, προβούμε σε διακρίσεις και δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να επιτρέπει να δίνονται διαφορετικά επιδόματα τέκνων στους εργαζομένους ανάλογα με το που ζουν τα παιδιά. Όταν οι γονείς τους πληρώνουν στο ίδιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ε, ή ε, τη φορολογία, δεν μπορούν να έχουν διαφορετικά επιδόματα τέκνων ανάλογα με το που ζουν τα παιδιά. Ε, είναι ανάλογα με τις εισφορές που πληρώνουν οι γονείς. Έχουμε το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και αυτή είναι και η στάση μα Όταν ερχόμαστε να αξιολογήσουμε ποιε είναι οι διάφορε προτάσει των κρατών μελών. Εγώ δεν μπορώ να προεξοφλήσω τι θα κάνουμε σε περίπτωση που θα δούμε τι θα γίνει στα διάφορα κράτη-μέλη και όταν γίνονται πράγματα τα οποία αντιτίθεται στην νομοθεσία θα αναλάβουμε πρωτοβουλία και θα αντιδράσουμε όπως το κάνουμε άλλωστε. κοινωνική ασφάλιση και ψηφιοποίηση. Όντως. Εμεί μπορεί να πάρουμε ό,τι πρωτοβουλία θέλουμε, να αξιοποιήσουμε και τα μέσα που έχουμε για να ελέγχουμε τα συστήματα και να ε, είναι όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Γι' αυτό ε, έχουμε αναπτύξει αυτή την πλατφόρμα ΕΣΥ και θέλουμε να ανασάρουμε και τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης έτσι ώστε και εκεί να μπούμε στην ψηφιακή εποχή και να κερδίσουμε για να φτάσουμε στους στόχους μας, αλλά με τρόπο ουσιαστικό. Σε ό,τι αφορά αυτό, τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν προσαρμοστεί μέχρι τα τέλη του 19. Είναι σαφές, είναι αποφασισμένο αυτό και για τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης απάντησα. Ε, προηγουμένως κύριε Μπάλας δεν είχατε έρθει ακόμα, δεν καταφέραμε να το παρουσιάσουμε ε, εγώ ήλπιζα να είναι στο πακέτο για τη δίκαιη μεταχείριση, το fairness package, αλλά δεν είναι τα τεχνικά δεδομένα ακόμα έτοιμα και δεν μπορούμε να κατεβάσουμε την πρόταση αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη, ε, ελεγμένη, δοκιμασμένη, γιατί οι κακές προτάσεις έχουν και κακά αποτελέσματα. Εργαζόμαστε όμως σε αυτό το τομέα. Για το Εράσμος, τριπλασιασμός των κονδυλίων, γιατί όχι τετραπλασιασμός. Ο καθένας γνωρίζει ότι είναι από τις βασικές μάρκες, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κόσμος το ξέρει, το εκτιμά και βοηθάει τους ανθρώπους να νιώθουν Ευρωπαίοι. Δίνει πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες σε πολλούς νέους, γι' αυτό θέλησαμε να το διευρύνουμε. Επίσης, αυτό τον καιρό Έχουμε και ένα εράσμους επαγγελματικό, εράσμους προ. Για, ε, προσεχώς θα ε, το παρουσιάσουμε αυτό για μαθητευόμενους στην επαγγελματική κατάρτιση και σε μαθητεία και κυρίως στα ε, πανεπιστήμια. θα πρέπει όλοι οι φοιτητές, οι σπουδαστές και τις τεχνικής εκπαίδευσης να μπορούν να συμμετέχουν. Ξέρουμε ότι είναι πενιχρά τα οικονομικά. Στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την επόμενη επταετία και μάλιστα ήταν ένα μικρό θαύμα που καταφέραμε να διπλασιάσουμε τον προπολογισμό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο, δεν μπορώ να αποφανθώ. Να πίεστε πάρα πολύ τα κράτη-μέλη σας, να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την Ευρώπη να έχουμε περισσότερα κονδύλια στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Τώρα δουλεύουμε με τα λεφτά που έχουμε. Και το Erasmus Plus διπλασιάζεται. Ας μην μειωθεί, να δούμε στο μέλλον αν μπορέσει να αυξηθεί. Για την απόσπαση των εργαζομένων. Χαίρομαι που θα συζητηθεί στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα. Είναι στην ημερήσια διάταξη. Μετά τον επιτυχή διάλογο. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, γι' αυτό. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να ψηφιστεί. Προσβλέπω στην υποστήριξη και στην πλειοψηφία. Έχει περάσει πολύ το Κοινοβούλιο την τελική πρόταση. Κύριε Μάν, σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά ταξίδια, άκουσα πολλά την τελευταία εβδομάδα. Πήρα και ε, μια επιστολή την οποία θα απαντήσω. Αλλά κάποιος που πάει ένα επαγγελματικό, σε ένα, ταξίδι, σε ε, ένα επαγγελματικό ταξίδι σε ένα κράτος μέλος ε, δεν είναι παροχή υπηρεσιών, δεν εμπίπτει στην απόσπαση των εργαζομένων θα απαντήσουμε στην επιστολή γραπτός για να γνωρίζουν και τα μέλη του Κοινοβουλίου που το ρώτησαν τι συμβαίνει και να είναι σαφή τα πράγματα. Για την Ελλάδα. Η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα, είναι γεγονός αυτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει προφανώ ότι δεν υπάρχουν πια υποχρεώσει. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν υποχρεώσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραμένει μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και κάθε άλλη χώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε λεπτομέρειε τι έχει συμφωνηθεί ακριβώ μεταξύ τη Ελλάδα και ε, των συναδέλφων μου αυτό που γνωρίζω είναι ότι όταν έγιναν τα νέα προγράμματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάναμε πρώτα μια μελέτη κοινωνικού αντικτύπου και πραγματικά είναι πάρα πολύ, ε, βελτιώθηκαν πολύ τα πιο επισφαλή ε, ε, προβλήματα, πιο επισφαλείς καταστάσεις. Σε θέματα εμπορίου ξέρουμε ότι γίνονται συμφωνίες, ε, υπάρχει πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Η συνάδελφος Ασίλια Μάλμστρομ νυχθημερών εργάζεται για να βρει την καλύτερη λύση κάθε φορά απέναντι σε μονομερές δηλώσεις και ενέργειες και ε, τα στρατηγικά μας συμφέροντα θα διαβιλεχθούν. Και μια ε, παρατήρηση για τη μη διάκριση. Έφυγε τώρα ο κύριος Μαρτά, αλλά θα του το διαβιβάσετε Έχετε απολύτως δίκιο όταν πρόκειται για τη διάκριση δεν λέμε ότι επιθυμούμε κάτι να γίνει, φυσικά το απαιτούμε να λυθεί. Εντάξει, επέλεξα λάθος λέξη να χρησιμοποιήσω. Και ζητώ συγγνώμη, δεν πρόκειται για επιθυμία, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Στην Ευρώπη δεν χωράνε διακρίσεις. Υπάρχει νομοθεσία που θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, πυκνή ε, παρέμβασή σας που έδωσε πολλές απαντήσεις. Ας περάσουμε στο θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης. Κάπως βέβαια έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Θα σας δώσω το λόγο ε, πάλι κυρία Επίτροπε για να κάνετε την εισαγωγή για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και μετά θα συνεχίσουμε με μια συζήτηση όσο γίνεται πιο πυκνή για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μετά στην ψηφοφορία. Μπορείτε να κάνετε μια σύντομη παρουσίαση. Ορίστε κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που με δέχεστε για να σας εξηγήσω την πρότασή μας περί αρχής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Πρόκειται για φιλόδοξη πρόταση που ως γνωρίζετε ωστόσο δεν είναι απομονωμένη ως πρωτοβουλία. Εντάσσεται στα πλαίσια μιας ε, ευρύτερης πολιτικής για την διασφάλιση δίκαιης πολιτικής με δίκαιους στόχους και τα είδαμε αυτά όταν ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνατε είναι στο κέντρο της προσπάθειας ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης και βέβαια και μαζί με τον κοινωνικό πυλώνα. Έχουμε αναλάβει διάφορες ε, ε, πρωτοβουλίες για να εξασφαλίσουμε τον δίκαιο χαρακτήρα της αγοράς εργασίας με κανονισμό για την πρόταση για την, ε, μάλλον με την οδηγία της απόσπασης εργαζομένων και μετά από μακρές διαπραγματεύσεις έχει μπει τώρα στην η διάταξη της επόμενης ε, Ολομέλειας. Επίσης Social Security Coordination που βρίσκεται τώρα σε συζήτηση στην Επιτροπή σας και όπου ελπίζουμε να αρχίσουμε τριμερείς διαλόγους στους επόμενους μήνες. Με αυτές τις πρωτοβουλίες, κυρία Πρόεδρε, θα έχουμε πλέον αναθεωρήσει τους οσιώδεις κανόνες Τη κινητικότητα τη εργασία. Το δε τελευταίο τμήμα που έχουμε θέσει επιτάπητο είναι πρόταση που θα διασφαλίζει ότι οι ουσιώδει αυτοί οι κανόνε εφαρμόζονται πραγματικά και ε, δεσμευτικά. Τα 70 εκατομμύρια Ευρωπαίων που ζουν και εργάζονται σε άλλη χώρα μέλη, μέλος, καθώς και πολλές επιχειρήσεις, αναμένουν από εμάς δικαιώματα και υποχρεώσεις που δεσπίζονται στο ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόζονται πραγματικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνει πραγματικότητα η δίκαιη ε, κινητικότητα των εργαζομένων πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι εθνικέ αρχέ να έχουν στα χέρια του όλου του μηχανισμού για να επιβάλλουν την τήρηση των προβλεπωμένων και πέραν των συνόρων, δηλαδή διαμεθοριακά. Δεν έχουμε πάντοτε πληροφορίε από του ομολόγου του. Οι, προφορίε προφορίες δεν είναι πάντοτε διαθέσιμες ή δεν διατίθενται. Δεν υπάρχει και γενικός μηχανισμός διαμεσολάβησης για όλα τα διαμεθοριακά θέματα. Για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Θα είναι διαρκής δομή που θα υποστηρίζει τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις και τους διακινούμενους εργαζόμενους. Η ELA θα καλύψει λοιπόν ένα πραγματικό κενό στην ε, επιβολή των κανόνων κινητικότητας και τα λοιπά και θα δώσει τους αναγκαίους μηχανισμούς για την ε, διάδοση της, ε, των πληροφοριών με τρόπο αποτελεσματικό. Λέω εγώ σαφώς, ποια πράγματα δεν θα κάνει η αρχή αυτή, θα είναι να αναλάβει δηλαδή τις, τα καθήκοντα των εθνικών αρχών. Ο σκοπό τη Ευρωπαϊκή Αρχή είναι να υποστηρίζει τι εθνικέ αρχέ για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου και όχι να τι υποκαταστήσει. Ο ELA λοιπόν δεν θα αλλάξει, η ELA μάλλον δεν θα αλλάξει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρων μελών. Το ίδιο δεν θα αναμειγνύεται με την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων που μπορούν να συμφωνούν στα πλαίσια των συστημάτων κοινωνικού διαλόγου των χωρών τους θα έχει επιχειρησιακό ρόλο να φροντίζει δηλαδή ώστε οι ευρωπαϊκοί κανόνες της κινητικότητας εργασίας να εφαρμόζονται με απλό, δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Η αρχή θα υποστηρίζει τις χώρες μέλη για θέματα διαμεθοριακής κινητικότητας κανόνες για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, ε, απόσπαση εργαζομένων, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και θα βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ χωρών μελών για να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές ε, επιπτώσεις της ε, κινητικότητας. Η πρότασή μας προβλέπει η αρχή να έχει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, να διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες ατόμων και εργοδοτών σχετικά με δικαιώματα και υποχρώσεις. Δεύτερο, να υποστηρίξει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών για την διαμεθοριακή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Νόμου και τρίτο, να προβλέπει διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις διαφορών, διαμεθοριακών διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών. Οι σκοποί αυτοί γίνονται πιο συγκεκριμένοι όταν εξετάσουμε και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που αναλαμβάνει η αρχή. Η αρχή θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα υπέρ των ατόμων και των εργοδοτών με διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ε, στην Αλοδαπή και βέβαια και με διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες. Χωρίς, να, ε, χωρίς επικάλυψη, αλλά με υποστήριξη των εφισταμένων συστημάτων και γι' αυτό προβλέπουμε η αρχή να χρησιμοποιεί τον πυλώνα URES και το Γραφείο Συντονισμού ΙΟΡΕΣ. και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και για την Ελβετία. Δεύτερο, η αρχή θα παρέχει επιχειρησιακή στήριξη στις εθνικές αρχές για να εξασφαλίζεται η αποκτηρισματική συνεργασία τους και αυτό είναι το βασικότερο καθήκον της αρχής εργασίας, Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Να φροντίζει δηλαδή για την ορθή εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κατά των καταχρήσεων. Θα διευκολύνει επίση τι ανταλλαγέ πληροφοριών μεταξύ εθνικών αρχών και θα συντονίζει και θα υποστηρίζει επιθεωρήσεις, δημοσιογραφικέ επιθεωρήσεις μετά από αίτηση των χωρών μελών ή μπορεί και να τι προτείνει η ίδια στι χώρε μέλη. Θα αναλάβει επίση το καθήκον διαμεσολάβηση μεταξύ των εθνικών αρχών σε περιπτώσει διαφορών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει επίσης ότι η αρχή θα συμβάλλει στο λεγόμενο capacity building των εθνικών αρχών, θα κάνει διαμεθοριακές αναλύσεις και αξιολογήσεις κινδύνων για θέματα διαμεθοριακής διακίνησης της ε, μάλλον, κυκλοφορίας της εργασίας και θα συνεννοείται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε περιπτώσεις που πρόκειται για μεγάλη κλίμακα αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Για την εκτέλεση όλων αυτών των καθηκόντων η αρχή θα βασιστεί στο έργο υφισταμένων οργανισμών Eurofund, SEDEFOP, EuroESA και EDF που είναι οι οργανισμοί που ε, δραστηριοποιούνται στο πεδίο των κοινωνικών θεμάτων και βέβαια συμπληρωματικά θα μπορούν να υπάρξουν συνέργειες βασισμένες σε εμπειρογνωμοσύνη, για παράδειγμα skills forecasting, η διαχείριση επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Θα συνεργάζεται και με άλλους συναρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως Ευρωπόλ και Ευρωτζάστ για θέματα αντιμετώπισης κλιματικών δράσεων στην, ε, στον χώρο της ε, ελεύθερης ε, κυκλοφορίας των εργαζόμενων. Άρα, οι προκλήσεις είναι σημαντικές και πολλές. Επίσης η δυσκολία του έργου είναι σημαντική, όμως σημαντική είναι και η αποφασιστικότητά μας να αποβεί επιτυχής η ίδρυση του, της ELA. ΕΕ. Με την ελευθερία διακίνηση των εργαζομένων, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε φιλόδοξοι. Η φιλοδοξία διακρίνει τις προτάσεις μας και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι και η κινητήρια δύναμη και για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία. Κατ' επανάληψη ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρία Πρόεδρε, πράγματι τόνισε την ανάγκη εφαρμογής, σωστής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ε, διαμεθοριακή κινητικότητα των εργαζομένων. Μιλώ για το ψήφισμα του 2016 για το κοινωνικό ντάμπινγκ και το 2014 για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως ε, στρατηγική για βελτίωση των ε, συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη. Αναμένω την ε, συμπαράστασή σας και βεβαίως είμαστε στην διάθεσή σας το προσωπικό μου γραφείο και εγώ, οι υπηρεσίες μας και εγώ να σας υποστηρίξουμε και εσάς βεβαίως και το Συμβούλιο Υπουργών στην νομοθετική διαδικασία. Με στόχο η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να είναι έτοιμη και λειτουργική το 2019. Ο ενθουσιασμός ε, του εισηγητού της ε, Επιτροπής σας θα παίξουν κρίσιμο ρόλο και των μελών σας βεβαίως και αναμένω με ενδιαφέρον τη συνεργασία μαζί σας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσουμε το λόγο στο ΕΛΚ. Ο κ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Τάισεν. Καταρχάς, που ήρθατε προσωπικά να μας κάνετε την παρουσίαση της πρότασης, αλλά και για την ίδια την πρόταση. Θέλουμε ένα περιβάλλον ειλικρινές, ε, χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό, ε, χωρίς εκμετάλλευση των εργαζομένων και οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι να προσπατεύονται σωστά. Και γιατί χρειάζεται αυτό, να είναι αυστηροί και ειλικρινείς κανόνες και στην περασμένη θητεία έγιναν πολλά και θα ψηφίσουμε για την οδηγία αυτή συντονισμός ε, κοινωνικής ασφάλισης, κινητικότητα στις μεταφορές, πολλά έγιναν. Αλλά οι καλοί κανόνες θα πρέπει να τηρούνται. Και τα τελευταία χρόνια οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι αυξήθηκαν όλο και περισσότεροι ε, πηγαίνουν να δουλέψουν από την άλλη μεριά των συνόρων. Είναι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι χρειάζονται επιθεωρήσεις ε, και η εξασφάλιση της στήριξης νομοθεσίας είναι κάτι που ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα. Άρα χρειάζεται διασυνοριακή συνεργασία και από εκεί ξεκινήσαμε για να κάνουμε αυτή την πρόταση την οποία και υποστηρίζω. Είμαι συγγητής στο Κοινοβούλιο, θα ασχοληθούμε με τους συναδέλφους και η πρόταση αποτελεί καλή βάση για συζήτηση. Το ιδανικό για μένα θα ήταν μια ε, αρχή εργασίας που να μην καλύπτει τα πάντα, αλλά να είναι αποτελεσματική σε αυτά που καλύπτει, στα λειτουργικά ε, στοιχεία ε, της υλοποίηση της της νομοθεσίας. Και χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αρχή που να έχει πολύ καλή περιγραφή του ρόλου της, αλλά να έχει και τα εφόδια εκείνα και τα πολεμοφόδια που χρειάζεται για να το επιβάλλει. Και θα ξέρω ότι γίνονται συζητήσεις στο Κοινοβούλιο για την παροχή ενημέρωση στους πολίτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι οπωσδήποτε ανάγκη να το κάνει συγκεκριμένη αρχή εργασίας. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό μάλλον το κοινωνικό δίκαιο και το εργατικό. Υπάρχουν και τα φορολογικά ζητήματα με διάφορες διμερείς συμφωνίες που έχουν ε, τα διάφορα κράτη-μέλη, Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αυτό πώς θα το αντιμετωπίσει. Ε, ε, μιλήσατε και για υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Πώς θα μπουν όλα αυτά κάτω από την ίδια ομπρέλα ας πούμε συμμετέχουν ε, στην εκπόνηση της πρότασης οι κοινωνικοί εταίροι επαρκώς. Μήπως χρειάζονται περισσότερα μέσα και εργαλεία για να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στις συνοριακές ε, επιθεωρήσεις και ελέγχους. Ε, μιλήσατε για συνεργασία με τη Europol. Στα σύνορα Βελγίου-Ολλανδίας έχουν πολύ θετικές εμπειρίες αυτό που θα το βάλετε σε μια σύντομη αναφορά, σε μια αιτιολογική σκέψη, δεν θέλουμε μια πιο συγκεκριμένη περιγραφή της συνεργασίας. Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής ε, εργασίας ε, στη μεσολάβηση, την οποία αναφέρατε μόνο επιγραμματικά. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα κληθούμε να τα απαντήσουμε το επόμενο διάστημα εδώ στην Επιτροπή μας. Σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να σας υποστηρίξω στο φιλόδοξο σχέδιό σας, το χρονικό δηλαδή, το 2019 να είναι έτοιμη και να λειτουργεί η αρχή αυτή και σε συνεργασία με εσάς, με το Συμβούλιο, αλλά κυρίως με τους συναδέλφους μου εδώ στην Επιτροπή. Θέλω να εργαστώ σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Σπυρίνσκι για το Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους διότι καταχράστηκα του χρόνου προηγουμένως. Δεν είχα επίγνωση του χρόνου που έτρεχε. Συνήθως δεν αμελώ το χρόνο. Βλέπετε δεν είχε αναφερθεί στην παρουσίαση του Αντιπροέδρου το θέμα. Αποτελματώνονται αμοιβέ ενώ έχουν εκτοξευθεί στα ουράνια ε, τα κέρδη και δεν έχουν καταβληθεί οι φόροι. Είναι τεράστιο θέμα που πρέπει να φωτιστεί. Όσον αφορά την αρχή εργασίας, έχω και εγώ την ίδια φιλοδοξία όπως οι συνάδελφοι και η κυρία Επίτροπος. Πρέπει να δημιουργήσουμε εύρυθμα λειτουργούς αρχή. Σχετικά με αυτό, να τονίσω τρία σημεία. Ένα που η ίδια η Επίτροπος ανέφερε, δηλαδή πρέπει να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών των κρατών μελών, η συνεργασία είναι ζωτική σημασία, πρέπει να βελτιωθεί. Ένα από τα ουσιαστικά προβλήματα όμω όσον αφορά τη δίκαιη κινητικότητα στην εσωτερική αγορά είναι η ανεπαρκή εφαρμογή των κανόνων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ε, που αφορούν τη διασυνοριακή κινητικότητα σε αυτό το πλαίσιο. Η αρχή πώ θα βοηθήσει, πώ θα συμβάλλει στην ενίσχυση των εξουσιών των εθνικών αρχών και των προνομίων αυτών σχετικά με αποτελεσματικότερου ελέγχου και πραγματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στι συνορικέ περιστάσεις συμπεριλαμβανομένων και σχετικών κυρώσεων ούτω ώστε να εφαρμοστούν στην πρακτική οι αρχέ τη κοινωνική δικαιοσύνη του πυλώνα. Δεύτερον, αν μία από ένα από τα καθήκοντα της αρχής είναι να βοηθά τις αρχές των κατών μελών για καλύτερη εφαρμογή των κανόνων και αρχών της δίκαιης κινητικότητας, δεν είναι σχετικό ότι οι περιπτώσεις παραβιάσεις της θετικής, της θεμητής κινητικότητας καθορίζονται σαφέστερα στον κανονισμό αυτό καθε αυτό. Και αναλυτική λειτουργία της αρχής που προβλέπεται αρκεί για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των διαφόρων διαφερομένων για την προστασία της ελευθερίας κινητικότητας. Δεν θα ήταν καλύτερο αν η αρχή ε, συναγάγει συμπεράσματα και εκδίδει ε, συστάσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη και τις αρχές σχετικά με τη στρέβλωση της αρχής της ενίας αγοράς, των αρχών της ενίας αγοράς όπως είναι η δίκαιη ανταγωνιστικότητα και η δίκαιη, ε, δίκαιος ανταγωνισμός. Και κάτι άλλο που σας ε, ενδιαφέρει από ό,τι ξέρω, προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιλύσει το πρόβλημα των πολλών δομών που ασχολούνται με την ε, κινητικότητα των εργαζομένων κάτι ευπρόσδεκτο. Και η απλούστευση πρέπει να ε, τονιστεί. Στο εγχείρημα δεν θα πρέπει να, να λησμονούμε τα σημαντικά καθήκοντα που εφαρμόζονται από δομές που θα απορροφηθούν από αυτή τη νέα αρχή. Σχετικά με αυτό, πώς η πλατφόρμα για τη μετώπιση αδήλωτης εργασίας θα διατηρηθεί εντός των πλησίων της αρχής. Η νέα αρχή δίνει δυνατότητα για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών για τη μετώπιση αδήλωτης εργασίας και να επερκεραστούν τα διάφορα προβλήματα και ελλείψεις και πιστεύω ότι αυτή η δυνατότητα που δεν είδε θα πρέπει να απολεστεί. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τρεμπέσιος τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και πάλι την Επίτροπο, την κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας παρουσιάσετε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με τον εκτενή και λεπτομεριακό τρόπο που το κάνατε. Βέβαια η πολιτική μου ομάδα και στο μέλλον θα εξακολουθεί να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Είμαστε όμως πεπισμένοι ότι η κατανομή των αρμοδιοτήτων όπως προκύπτει από, την Ευρωπαϊκή, από τις συνθήκες θα πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί. Και ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας δεν θα έχει επιπλέον αρμοδιότητες, θα περιοριστεί ε, στα θέματα της και θα διαφυλαχθούν και αρμοδιότητες των κρατών μελών για να μπορέσει να έχει μια προστιθέμενη αξία αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, κατά την άποψή μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να λειτουργεί ως αρχή που θα υποστηρίζει και θα συμπληρώνει τα κράτη-μέλη χωρίς να τα υποκαθιστά για τις αναλύσεις της αγοράς εργασίας, για τη συνεργασία, για την ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών, για την ε, δημιουργία ικανοτήτων, το capacity building και την υποστήριξη, ε, θα έχει μεγάλο όφαλος η ανταλλαγή πληροφοριών είναι χρήσιμη για την καταπολέμηση της κοινωνικής απάτης, αλλά προσοχή, υπάρχουν κίνδυνοι όταν συγκεντρωτικά συλλέγονται στοιχεία. Ε, οι μεγάλες οργανώσεις είναι βάλωτες ε, στο ε, ε, έγκλημα το ηλεκτρονικό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή συγκεντρωτικών στοιχείων. Σε ένα σημείο που δεν αναφερθήκατε καθόλου, αλλά είναι πολύ σημαντικό για μας και για την πολιτική μου ομάδα, το ECR έχει δυσκολίες, είναι η χρηματοδότηση αυτής της υποσύσταση αρχής. Αυτό αφορά από τη μια τα έξοδα του οργανισμού του ίδιου τα λειτουργικά και το δεύτερο πόθεν Πού θα τα βρούμε. Ξέρετε ότι έρχεται το Brexit και ο πίτροπος Σότιγκερ ε, παρουσίασε το νέο προπολογισμό, αλλά παραμένουν οι ε, αγωνίες και αβεβαιότητες για τη χρηματοδότηση. Ειδικά η πολιτική μου ομάδα ε, έχει λάβα τη στη μεγάλη δημοσιονομική πειθαρχία θα πρέπει να ε, κοιτάξουμε αν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν χρειάζεται να συνεχιστούν και να βρεθούν από εκεί κάποια αναπορόφητα κονδύλια από τις ε, γραμμές αυτές του προπολογισμού για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί αυτή η αρχή. Θα χαιρόμουν να αναφέρω σας τα λίγο και σε αυτό το σκέλος χρηματοδότησης. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την πρότασή σας άλλο ένα κομμάτι στο όλο ένιγμα για να έχουμε σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά την αναθεώρηση του ζητήματος της απόσπασης, ε, της κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Είπατε ίδια και διάβασα κιόλα ότι ο ρόλος της νέας αυτής υπηρεσίας εργασίας θα είναι να εφαρμόσετε αποτελεσματικά το κοινοτικό δίκαιο και να απεφευθούν καταχρήσεις και απάτη. Βλέποντας τα καθήκοντα τους κανόνες, το ρόλο κλπ. του ELA, αυτού του φορέα. Θεωρώ ότι οι δεσμεύσεις είναι πολύ σημαντικές που αναλαμβάνονται και το έργο της αρχής. Όσον αφορά την πρόταση, το ELA θα αντικαταστήσει κάποιες υφιστάμενες δομές. Επίσης θα έχει τη διαχείριση του EURES και πρέπει να συνεργάζεται με πολλούς φορείς, αρμόδιες αρχές κλπ. Έτσι δε περαιτέρω αναφέρεται ότι αν εντοπίσει κάποιες ατασταλίες εκτός του πεδίου που καλύπτει όπως στον τομέα υγείας και ασφάλειας θα πρέπει να αναφέρει αυτές τις περιπτώσεις και να συνεργάζεται εν τη αυτή περιπτώση με τις αρμόδιες αρχές. Η ερώτησή μου δοθέντος του αριθμού των φορέων που θα αντικατασταθούν από την υπηρεσία. Και χιλιάδες φορείς με τους οποίους θα πρέπει να συνεργάζεται ο ELA. Άρα η εντολή του είναι πολύ σημαντική. Πιστεύετε ότι ο προϋπολογισμός που προτείνατε αρκεί? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη. Ετέθη από τον κύριο Λέντας και από τον κύριο Πυρίνσκι εν μέρη το ερώτημά μου. Πώς. Αναφέρθηκα στην υγεία και ασφάλεια. Αν η υπηρεσία αυτή εργασίας, η LA, έχει ένα ρόλο εκτός του πεδίου της αρμοδιότητάς της. Αν εντοπίσει κάτι πρέπει να το αναφέρει και να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές. Τι διάβλους χρησιμοποιεί. Οι προθέσεις καλές και αγαθές αλλά χρειάζονται λεπτομέρειες για το πώς θα εφαρμοστούν κάποια πράγματα. Τέλος. Σχόλιο. Βλέποντας το έργο του ELA, προφανώς πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργεί ο φορέας επαρκώς, σωστά. Πώς. Πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα απ' όλα ότι το ESSI θα λειτουργεί ο κ. Μπάλλα ήδη το ρώτησε το θέμα. Δηλαδή κατά πόσο τα κράτη-μέλη θα έχουν το σύστημα αυτό έτοιμο μέχρι το 2019. Η απάντηση σας ήταν ότι θα έπρεπε. Ερώτηση. Από ό,τι γνωρίζετε, αυτά που ξέρετε τώρα, πιστεύετε ότι θα το εφαρμόσουν τα κάτι μέλη και αν όχι όλα τα κάτι μέλη τουλάχιστον ένα σημαντικό ποσοστό των κρατών μελών θα συμμορφωθεί και θα τα εφαρμόσει όλα αυτά όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Γκουε. Η κυρία Λόπες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Επίτροπε, πολύ για την πρόταση που μα ε, παρουσιάσατε σήμερα το πρωί. Γενικώ, είμαστε θετική απέναντι στην πρόταση να συσταθεί Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αν στόχο έχει την καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ και την εργασιακή απάτη. Για να λειτουργεί η εσωτερική αγορά θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο και με ίσο τρόπο να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες. Οπότε αξιολογούμε θετικά όλες τις πρωτοβουλίες που μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και το συντονισμό των εθνικών αρχών. Τι συμβαίνει όμως τώρα. Δυστυχώς διαπιστώνουμε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη παραβιάζουν κάθε μηχανισμό ε, ελέγχου και παρακολούθησης και του κοινοτικού εκτιμένου. Γι' αυτό η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι αυτή αξιέπαινος ο στόχος κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ, αλλά φοβάμαι ότι ε, μπορεί να μείνει κενό περιεχομένου ε, σχέδιο χωρίς καμία δυνατότητα αντίδρασης για να επιβάλλει τους στόχους τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που ε, σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία κάνει προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ε, τερματιστεί αυτή η μάστιγα. Και όταν έρθει η ώρα της αλήθειας μηδένει στο πηλίκο. Το είδαμε και με τη νέα νομοθεσία για την απόσπαση των εργαζομένων και πάλι βλέπουμε διαφορετική αμοιβή για την ίδια εργασία. Ερωτώ λοιπόν και διερωτώ με ειλικρινά θα βοηθήσει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να καταπολεμηθεί το ντάμπινγκ και οι καταχρήσεις. Ενώ οι ίδιοι κανόνες που θα πρέπει να είναι θεματοφύλακας αυτών δυστυχών δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η κριτική έρχεται να θυμίσει τη σημασία που έχει ε, η καταπολέμηση και η πάταξη του κοινωνικού ντάμπινγκ. Με αυτό θα πρέπει να ασχοληθεί. Ο συντονισμός των εθνικών αρχών θα πρέπει να γίνει με την απλή λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σωστή ερμηνεία της νομοθεσίας που αφορά όλους τους εργαζομένους. Δεν είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι για τον τρόπο με τον οποίο ο νέος αυτός οργανισμός θα καταφέρει να συντονίσει καλύτερα, ουσιαστικά καλύτερα, ε, με ποιους μηχανισμούς και τι μηχανισμούς διαθέτει ε, για να ενεργεί σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων και μη σεβασμού αυτών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ράνκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε. Η πρότασή σας παραδέχεται την πραγματικότητα που γνωρίζαμε επί μακρόν ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Άρα συνάχει, χρειάζεται και υποπτική αρχή για να εξετάζει αυτά που συμβαίνουν στην αγορά εργασίας. Καταρχήν, άκρος ευπρόσδεκτη η πρότασή σας. Στο τέλος όμως οι διατάξεις είναι πολύ περίπλοκες, αλλά η πολιτική αφορά δύο πράγματα πολύ συχνά, εξουσία και χρήμα. Και αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθούν και ερωτήσει μου. Βλέποντας την πρότασή σας, είναι πολύ ενθαρρυντική. Έχει τεθεί θετικότατα. Ε, Διαμεσολαβεί, διευκολύνει κλπ. Ερώτηση. Στο τέλος η αρχή θα έχει πραγματικά εξουσία. Τι συμβαίνει σε περίπτωση σύγκρουσης. Θα μπορεί να πιέσει τα κράτη-μέλη αυτή η αρχή, ούτω ώστε να παράσχουν κάποιες πληροφορίε εντό χρονικού διαστήματος που είναι απαραίτητο για να υπάρξει δράση σε περίπτωση παράβασης και κατάχρηση. Αυτό συνέβη τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι Δεν πρέπει να υπάρχει απλή βούληση συνεργασία των εθνικών φορέων, τι ε, εργασία, επιθεώρηση εργασία συνεργαστούν, αλλά τι εξουσία θα έχει αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή. Μετά χρήματα. Μιλήσατε για, για κοινού ελέγχου που θα κοστίζουν. Πόσα χρήματα. Πόσοι έλεγχοι θα γίνουν. Πώς εξασφαλίζεται ότι θα παρασχεθούν τα χρήματα, ότι θα υπάρχουν εναγκαίοι πόροι για να γίνει αυτό. Πολύ κρίσιμο αυτό. Ο ΕΛΑ θα πρέπει να λειτουργεί, αλλά να έχει και μια επιρροή, πραγματική επιρροή στην αγορά εργασία. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ, κυρία Άνκη, για αυτό που είπατε. EFTD. Αν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος του EFTD, όχι. Κάποιος εκπρόσωπος του ENF, όχι. Πάμε στην κυρία Χέλγα Στίβενς που έχει ζητήσει το λόγο και έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, γνωρίζετε ότι σας υποστηρίζω απολύτως ε, ε, στην προσπάθειά σας να καταπολεμήσετε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Ε, εδώ είναι θύματα εργαζόμενοι σήμερα και οι ντόπιοι και οι μετακινούμενοι αποσπασμένοι. Είναι ένα καλό βήμα λοιπόν για τη διασυνοριακή απάτη για να τερματιστούν αυτές οι αθέμητες πρακτικές. Ωστόσο έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες επιφυλάξεις ε, στην πρότασή σας για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Πρώτον, θέλω να τονίσω ότι η αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι να κάνουν τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Και οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας έχουν κάθε μια το δικό τους τρόπο εργασίας. Εγώ ανησυχώ μήπως η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έρχεται να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σήμερα, αλλά αύριο υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει. Χρειάζεται μια αξιολόγηση. Ε, σε, ε, σε περίπτωση πούμε, που δεν λειτουργεί καλά η Ευρωπαϊκή Αρχή, τι θα γίνει. Διαβάζω στην πρόταση ότι μετά από μία πενταετία θα αξιολογηθεί αν θα πρέπει ή να αλλάξει η εντολή του οργανισμού αυτού. Φοβούμε όμως ότι σήμερα θα ε, γίνουν τα πρώτα βήματα για μια πανευρωπαϊκή επιθεώρηση εργασίας. Μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι δεν έχετε αυτή την πρόθεση. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία. όχι να παίρνει όλο και περισσότερε αρμοδιότητε και εξουσίε από τα κράτη-μέλη. Δεύτερη σύντομη ερώτηση. Μπορείτε να με ενημερώσετε για το νομικό καθεστώ τη Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Για παράδειγμα, ποιε είναι οι σχέσει της με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Περιμένω τις αποφα... Ε, απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'll give the... Ευχαριστώ. Ο κ. Τέτσον, έχετε το λόγο. Ο Ζαν Κλώτ παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λέγοντας τα εξής είναι παράλογο μια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή να επιτηρεί κατά πόσο τηρούνται τα τραπεζικά στάνταρ και να μην υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας που να φροντίζει να υπάρχει δικαιοσύνη στο εσωτερικό της ευρωπαϊκής αγοράς και θα τη δημιουργήσουμε αυτή την αρχή. Και εμεί θέλουμε μια δίκαιη εσωτερική αγορά αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργεί τόσο σωστά. Εκεί που έχουμε διασυνοριακές μορφές απασχόλησης ε, χρειάζεται και ε, να υπάρχουν διασυνοριακοί έλεγχοι. Οι κοινωνικές προδιαγραφές ταλαιπωρούνται από εταιρείε θηρίδες ε, και τελικά είναι εις βάρος των εργαζομένων να παίζει και τις ε, νομοταγείς εταιρείε που τηρούν τα πρότυπα και τις προδιαγραφές ε, και το εργατικό δίκαιο. Ρωτώ λοιπόν, αν κατάλαβα καλά κυρία Επίτροπε, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπεται να γίνονται μόνο επιθεωρήσεις εργασίας που θα ζητεί εκάστοτε χώρα. Και όταν γίνονται αυτοί οι έλεγχοι, τι θα γίνει. Δεν είναι σήμαντο να έχουν το δικαίωμα και οι κοινωνικοί εταίροι να ζητούν τους ελέγχους, όχι μόνο τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να γίνονται πραγματικά επιθεωρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι επί τόπου οι κοινωνικοί εταίροι γνωρίζουν καλύτερα πώς έχει η κατάσταση στη χώρα και μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα αν υπάρχουν κάποιες παραβάσεις και παραβιάσεις των κοινωνικών και εργασιακών ε, προδιαγραφών. Τι πιστεύετε για την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιόγκες και μετά <clears throat> η κυρία Τάισιν για να απαντήσει. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα καθυστερήσουμε λίγο με την ψηφοφορία, με την έναρξη ψηφοφορίας. Αλλά είναι σημαντικό θέμα. Άρα μην ανησυχείτε. Πρώτα η κυρία Γιονγκέριος και μετά η κυρία Τάση. Θα είμαι σύντομη. Ε, δεν θα ε, χάσω χρόνο με το να σας πω πόσο πολύ χαίρομαι για την πρόταση. Δύο ερωτήσεις. Γιατί δεν υποχρεώνει η Επιτροπή της Εθνικές Επιθεωρήσεις να συμμετέχουν. Αυτό είναι το ένα. Στι επιθεωρήσει. Δεύτερο. Δεύτερη ερώτηση. Αν υπάρχει μια ξεκάθαρη περίπτωση εκμετάλλευσης. Αυτές οι υποθέσεις πώς θα αχθούν ενώπιον του, της ELA. Τα συνδικάτα θα έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλουν συγκεκριμένες υποθέσεις και πόσο γρήγορα θα ανταποκρίνεται η ELA. Τελευταία ερώτηση. Θα υπάρξει εν τέλει ένας μαύρος κατάλογος των επιχειρήσεων, ας πούμε, ε, ε, γραμματοκιβωτίου, οι οποίες καταχρώνται του συστήματος. Διότι νομίζω <clears throat> ότι κάτι τέτοιο πράγματι θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο πάλι στην ε, Μάριαν Τάισεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη, ξέρω ότι επήγεστε να κάνετε την ψηφοφορία και ίσως και μετά να αποχωρήσετε και από τις Βρυξέλλες. Πρώτα, Γερούν Λέναρτς. Γερούν καλή τύχη και καλή επιτυχία. Στην έκθεση είναι βαριά αυτή η αποστολή. Πάντως φαίνεται ότι έχετε μεγάλη φιλοδοξία να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια και να ε, γίνει λειτουργική αυτή η αρχή. Γιατί τελικά το αποτέλεσμα μετράει και εκ του αποτελέσματος ε, θα κρυθούμε να δούμε πώς θα προχωρήσει, πώς θα αρχίσει να λειτουργεί και τι θα αποδώσει αυτή η αρχή. Κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας ε, ρώτησες πολλά πράγματα, δεν θα μπω στην ουσία, ήταν πολύ εύστοχες οι ερωτήσεις όσο και οι παρατηρήσεις θα το, το μελετήσουμε και οι νομοθέτες. Πρέπει προσβλέπω στη συνεργασία μας και ε, στην τελική πρόταση του Κοινοβουλίου. Καλή επιτυχία και οι συγγητέ και τα μέλη του Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα για να το μελετήσουν σε βάθος και όσο γίνεται ε, να βελτιώσουν την πρότασή μα όπως πάντα γίνεται. η παρουσίαση αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή, εμπεριστατωμένη, την υποστηρίζει όλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την έχουμε μελετήσει, την έχουμε δουλέψει. Ε, βεβαίως πάντα χωρούν ε, βελτιώσει με χαρά να γίνει, όπω και σε άλλα θέματα. Ε, άλλη ερώτηση. Μια ερώτηση που επανέρχεται ξανά και ξανά, κυρία Πρόεδρε. Για ποιο λόγο δεν υποχρεώνονται να συνεργαστούν τα κράτη-μέλη και όταν ε, δείχνουν προθυμία να το κάνουν αυτό στα πλαίσια της ΕΛΑ, τι θα κάνουμε, θα επιβάλλουμε κυρώσεις. Τα κράτη-μέλη έχουν κάποιες υποχρεώσεις ε, ε, που ορίζονται από την νομοθεσία, από την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων Υπάρχουν στο σχετικό κανονισμό για το συντονισμό των, συστημάτων εθνικ... Ε, εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το 2014 ψηφίσατε μια πρόταση οδηγίας κτλ. Ε, αυτά ορίζονται από την νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία τι κάνει. Φροντίζει ε, ε, κάποιες υπηρεσίες να συνεργάζονται με συνδέσμους ε, υπαλλήλου από τα κράτη-μέλη σε μια επιχειρησιακή δομή μόνιμου χαρακτήρα σε έναν οργανισμό για να υποστηρίζει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτά τα πράγματα. Εμείς θεωρούμε ότι η εμπιστοσύνη εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική και η πίεση θα αυξηθεί. Όταν καθημερινά συνεργάζονται άνθρωποι από επιθεωρήσει εργασία και είναι στα ίδια γραφεία, στον ίδιο διάδρομο και βλέπονται καθημερινά, έτσι θα υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη ενθάρρυνση έτσι ώστε να ανταλλάσσουν και πληροφορίε αυτέ που ζητούνται και να λένε στα κράτη-μέλη τι πρέπει να κάνουν για να κάνουν ελέγχους και επιθεωρήσεις για να ε, καταπολεμούν την απάτη και το κοινωνικό ντάμπινγκ. Λοιπόν, είναι θέμα συνεργασίας και οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών, ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση. Φυσικά, άμα δεν κάνουμε τίποτα, έχουμε ε, στην νομοθεσία προβλέπονται και κυρώσει για να προχωρήσουμε. Για την πλατφόρμα, την ηλεκτρονική κατά της μαύρης εργασίας, αδήλωτης κλπ αυτό υιοθετείται και ενισχύεται. Είναι καλή αυτή η πλατφόρμα, λειτουργεί, αποδίδει και θα ενταχθεί ε, στην Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας έτσι ώστε να έχουν ακόμα περισσότερα εργαλεία ε, στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι. Δεν καταργείται αυτή η πλατφόρμα, εντάσσεται στην ΕΛΑ. Παραμένει αυτό το, αυτή η μονάδα, αλλά σε άλλη δομή. Για τη χρηματοδότηση κοιτάξαμε πάρα πολύ, μελετήσαμε τι χρειαζόμαστε, βέβαια πάντα με αποτελεσματικότητα. Ξέρουμε πόσοι υπάλληλοι χρειάζονται, ε, ποια είναι η χρηματοδότηση, έχει κοστολογηθεί, έχει προϋπολογιστεί και εγγραφεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προβλέπονται τα αντίστοιχα κονδύλια και ο προϋπολογισμός, ένα δις, ε, όλοι αυτοί οι υπολογισμοί έχουν ελεγχθεί από τους αρμοδίους για τα οικονομικά. Και είναι αρκετός ο προϋπολογισμός. Τι θα κάνουμε αν παρόλα αυτά παραμείνει το κοινωνικό ντάμπινγκ, έλεγχος και σε περίπτωση παραβίαση, παράβαση νομοθεσία. Υπάρχουν οι συνήθει διαδικασίε προσφυγή, επί παραβάση κτλ. Τα λέει αυτά η νομοθεσία. Προβλέπονται, φυσικά τα έχουμε σκεφτεί. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία τι κάνει, επιθεωρήσει, ελέγχου, συντονισμό. Αυτό είναι ο ρόλο τη και το έργο τη. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αναγκαίο. Κάτι που ρώτησε η κυρία Χάρκινγκ. είναι κατάλληλο ο προπολογισμό, όλα αυτά έχουν προβλεφθεί και συμπεριληφθεί στο PDP και στου επόμενου ε, προπολογισμού. Πώς θα τα ελοπίσουμε όλα αυτά. Γιατί καλές οι προθέσεις, αλλά θα πρέπει να είναι ε, σωστή και η δομή και να υπάρχει και κάποια κρίσιμη μάζα αιτήσεων. Γι' αυτό συστήσαμε μια ομάδα συμβουλευτική όπου συμμετέχει σε τεχνικό επίπεδο και κάποιος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνεδριάσει μία φορά. Δηλαδή τώρα συζητούμε ήδη τον τρόπο με τον οποίο θα στηθούν όλα αυτά και θα ορθοποδήσουν. Γιατί Καλό είναι να κάνεις μια νομοθεσία, αλλά μετά θα πρέπει να το στήσεις και τον οργανισμό. Τώρα αυτό μας απασχολεί. Ακόμα πριν την νομοθετική διαδικασία, πριν την ολοκλήρωση της δηλαδή, κοιτάζουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, ακούμε τον καθένα, έτσι ώστε να, στηθεί σωστά από την αρχή αυτός ο μηχανισμός και αυτός ο οργανισμός για να αναλάβει το έργο που του αναλογεί. Ε, για το, η πλατφόρμα ESI, η SSI, θα πρέπει από το 2019 να το υλοποιήσουν αυτό το κράτη-μέλη. Τους το θυμίζουμε συχνά ε, όταν ε, πλησιάζει η ε, θέση σε ισχύ ενός νόμου. Θυμίζουμε στα κράτη-μέλη ότι έχουν κάποιες υποχρεώσεις και συνεργάζονται. Έγιναν πολλές ερωτήσεις γιατί προχώρησα παραπάνω, δεν έχουμε αρκετούς επιθεωρητές. Πόσους υπηθεωρητές θα έχουμε ακριβώς εκεί, σε αυτόν τον οργανισμό και ποιος θα κάνει τι. Καλά, θα τα δούμε αυτά όταν στηθεί ο οργανισμός. Σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας βρισκόμαστε τώρα. Κατά τα άλλα, για το προσωπικό προβλέπονται τα κονδύλια στην πρόταση και όπως σας είπα είναι αρκετά και είναι και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχει συνυπολογιστεί, όχι μόνο για τον ε, προπολογισμό οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ζητούν ελέγχους. Βεβαίως, προφανώς. Αλλά αυτό είναι θέμα εθνικού επίπεδου, όχι ευρωπαϊκού. Έχουμε μια ομάδα ενδιαφερομένων που εργάζεται και οι stakeholders και συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι και τα συνδικάτα και μπορούν και δι' αυτού του τρόπου να το κάνουν, αλλά βασικά είναι θέμα κράτους μέλους. Θα πρέπει να ζητούν ελέγχους από τις εθνικές αρχές και επιθεωρήσεις. Ορισμένοι θεωρούν ότι είναι δούριος ύπος αυτή η αρχή για να αφαιρέσουμε αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Θέλουμε να ενισχύσουμε τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις ομάδες των επιθεωρητών και ελεγκτών για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Δεν αφαιρούμε ε, από τα κράτη-μέλη την εξουσία αυτή. Δεν φτιάχνουμε ευρωστρατό επιθεωρητών εργασίας. Υπάρχει και ρήτρα αναθεώρησης και αυτό είναι ένα στοιχείο καλής ε, πρακτική και διαχείριση. Όταν κάνει μια νομοθεσία και δημιουργεί ένα όργανο, θα πρέπει να δει μετά από ένα διάστημα πώ λειτουργούν, αν αποδίδουν και μετά να αξιολογεί και αν χρειαστεί να αλλάζει και κάποια πράγματα. Επίσης θέλω να πω ότι η αρχή της επικουρικότητας και της αναλογικότητας βεβαίως βρίσκουν εφαρμογή και εδώ. Αυτό το κάνουμε στην πρότασή μας. Προχωρούμε τόσο όσο να μην μπαίνουμε σε χωράφια επικουρικότητας και αναλογικότητας. Δεν πρόκειται να αναλάβει τίποτα. η επιθεωρήσεις εργασίας βεβαίως είναι ε, εθνική υπόθεση. Δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή αρχή να πάει σε μια χώρα και να πει καλημέρα σας από σήμερα να λαμβάνω εγώ τους ελέγχους. Θα πρέπει να συνεργάζονται οι επιθεωρήσεις και να υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή αυτή αρχή. Και με υλικό και με υποδομή και με ενημέρωση από συναδέλφους σε άλλη χώρα για να διευκολύνουν, να έχουν την, την επιμελητία, την υποστήριξη, την τεχνική και συντονισμό ενδεχομένω επιθεωρήσεων που γίνονται ταυτόχρονα οι έλεγχοι σε διάφορα κράτη-μέλη. μαύρος κατάλογος εταιριών. Δεν ξέρω, δεν προβλέπεται στην νομοθεσία μας. Στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα ε, λειτουργήσει συγκεκριμένα η ΕΛΑ. Αλλά αυτό έχουν νόημα σε εθνικό επίπεδο, όχι σε ευρωπαϊκό. Πρόεδρε, ελπίζω να απάντησα όσο μπορούσα στο χρόνο που μου δώσατε. Πάντω, ένα είναι γεγονό. δεν είναι τελευταία φορά που θα συζητούμε αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντική πρόταση και εύχομαι στα μέλη του Κοινοβουλίου καλή επιτυχία στι εργασίε και ελπίζω από κοινού να φέρουμε σε πέρας αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Τάισεν που περάσατε το χρόνο αυτό μαζί μας και απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις, προσπαθήσατε τουλάχιστον. Προς ενημέρωσή σας, αμέσως μετά την ψηφοφορία, σε ένα τέταρτο περίπου, ε, έχουμε ένα εργαστήριο για τη δημιουργία αυτής της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής ε, Εργασίας. Ελπίζω να παραμείνετε αμέσως μετά την ψηφοφορία. Θα έρθουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μας βοηθήσουν σε αυτό το εργαστήριο. Δεύτερον, προς ενημέρωσης, η ψηφοφορία για την απόσπαση των εργαζομένων θα λάβει χώρα την τρίτη της επόμενης εβδομάδος στο Στρασβούργο το πρωί. 9-10 η ώρα νομίζω το πρωί. Εστε παρόντες, παρακαλώ συμμετάσχετε στην ψηφοφορία. Τούτων λεχθέντων θα ψάξουμε να βρούμε τις κάρτες ε, ψηφοφορίας. Ξεκινάμε την ψηφοφορία, φίλοι μου. Θα έχετε, πιστεύω, βάλει τις κάρτες σας ε, στα μηχανήματα. Θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, συμβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμπλήρωμα 1, υπέρ. Κατά αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται ο έλεγχος. Άρχισε δεν άρχισε. Δεν δουλεύει το δικό μου το μηχάνημα. Α, ωραία δουλεύει. Βοήθησε το χτυπηματάκι αυτό. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 υπέρ, 16 κατά. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προσθήκη 2 να ζητήσω ονομαστική ψηφοφορία ακούγεται από κάτω Πρόεδρος ονομαστική ψηφοφορία για το συμπλήρωμα 2 υπέρ λέει πρόεδρος κατά Ξανά ονομαστική. Ψηφίζουμε, λέει η Πρόεδρος. Θα ψηφίσουμε για την ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία απλώς. Δεκατέσσερις χρειάζονται. Έντεκα μέλη. πάνω από 11 μέλη. Μπορείτε να καθίσετε. Λοιπόν, για το συμπλήρωμα 2 ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ 14 κατά και 2 αποχές. Πάμε στη συμβιβαστική 4 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμπλήρωμα 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμπλήρωμα 4. Υπέρ. Κατά. Για την προστίκη 4 ψηφίζουμε. Ξεκινάει τώρα. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προστίκη 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για την προσθήκη 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Προσθήκη 6. Λοιπόν, υπέρ της προσθήκης 6, παρακαλώ. Μάλλον ονομαστική ψηφοφορία η οποία άρχεται τώρα για την προσθήκη 6. Πέρας για την προσθήκη 6. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. Προσθήκη 7. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προσθήκη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προσθήκη 9 υπέρ κατά έλεγχος ή την προσθήκη 9 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 ψήφοι υπέρ, 13 ψήφοι εναντίον. Ονομαστική ψηφορία για το 10 και 11 παρακαλώ. Ακούγεται από κάτω. Για τη 10 και 11. Για την προστίκη 10 θέλετε ονομαστική ψηφοφορία. Καλώς. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την προστίκη 10 συγγνώμη πέρας για την προσθήκη 10 εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ 13 ψήφους εναντίον προσθήκη 11 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται πέρας εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ 14 ψήφους εναντίον και 2 αποχές. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συνεισφορά της Επιτροπής στο διαθρωμένο διάλογο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους εναντίον και καμία αποχή. Ευχαριστώ. Άρα προχωρούμε. workshop το εργαστήριο το εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας συνεχίζει η Πρόεδρος Κοιτάξτε, θα σας δώσω δύο λεπτά για να μπορέσετε να αποχωρήσετε και μετά θα συνεχίσουμε. Okay, then we... Η πρόεδρος. Καλά, λοιπόν, ας αρχίσουμε με το εργαστήρι. Δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Έχουμε κοντά μας τον Ντένις Λέγκτον, που είναι από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ευχαριστώ θα του δώσω το λόγο ξαναλέω το όνομά του Γκέντεν. Τον ευχαριστώ. Κάθεστε καλά εκεί που είστε ή προτιμάτε να έρθετε εδώ μπροστά. Ναι, ναι, αν είναι δυνατόν, ναι, ναι, ορίστε, ελάτε. Κοπιάστε. Ώστε να μπορούν να σας βλέπουν καλύτερα και τα μέλη. Επίσης, η κυρία Αλεξία Μανιάκα Γρίβα παρακαλείται και αυτή να έλθει να καθίσει εδώ. Ευχαριστώ, πολύ κύριε Γκέντεν για την παρουσία σας εδώ και ε, κάθεστε ώστε να σας βλέπουν όλοι. και βεβαίως παρακολουθούν και ε, κάποιοι από τους υπολογιστές στα γραφεία τους. Θα σας δώσω το λόγο για να εξηγήσετε τη μελέτη αντικτύπου για την ε, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση που απευθύνατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντικαθιστώ τον κύριο Βαντών, λέγομαι Πανκάλντι και όχι Κέντεν. Ε, βλέπετε και στη διαφάνεια. Θα πω με λίγα λόγια ποια είναι η μελέτη αντικτύπου και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ασχοληθήκαμε με τέσσερα βασικά θέματα, προβλήματα, τι επιθυμούμε να επιτύχουμε, τα καθήκοντα που θα αναλάβει η LA και τέλος πώς θα τα εκτελέσει τα καθήκοντα αυτά. Θα εξηγήσω τα διάφορα αυτά θέματα και αν θέλετε να αρχίσουμε με τα προβλήματα που έχουμε, εμείς έχουμε εντοπίσει δύο ιδίως. Το πρώτο είναι ανεπαρκείς πληροφορίες για τους πολίτες, ε, για ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν, επίσης για τους εργοδότες και βέβαια και η διοικητική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που υποτίθεται ότι επιβάλλουν την τήρηση των κανόνων. Τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα πιο συγκεκριμένα. Τα βλέπουμε στη διαφάνεια εδώ που επιγράφεται problem drivers. Δεν είναι αχαρτογράφητα τα εδάφια αυτά. Υπάρχουν διοικητικές πρακτικές που αντιμετωπίζουν τα επιμέρους προβλήματα. Ωστόσο, για κάθε ένα από τα καθήκοντα που ανέπτυξε πριν η κυρία Τέισεν, υπάρχει έλλειψη συστημικότητας. Υπάρχει έλλειψη στήριξης επαρκούς στελεχικού δυναμικού ή εφαρμογής στους διάφορους τομείς. Και αυτά είναι που έχουμε εντοπίσει. Αφενός βλέπουμε ανεπαρκείς ή ατελείς πληροφορίες. Από την άλλη μεριά Έχουμε όλα όσα έχουν να κάνουν με διοικητική συνεργασία. Πάλι εδώ ατελή η ανεπαρκή ικανότητα. Έχουμε ε, συστήματα πληροφορικής, συστήματα της ε, security coordination, αλλά υπάρχει διαρκής ανάγκη επικαιροποίησης και ε, συνεργασίας των συστημάτων αυτών. Επίσης η ικανότητα οργάνωσης της συνεργασίας. Εδώ υπάρχει ιδίως έλλειψη κοινών διαδικασιών. Υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες μεταξύ χωρών μελών. Υπάρχουν και φόρουμ σε διεθνές επίπεδο, αλλά αυτά όλα συναποτελούν μέρος διμερών συμφωνιών μεταξύ επιμέρους χωρών μελών και δεν είναι πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. Το δε ίδιο συμβαίνει και για τους μηχανισμούς για κοινέ δράσεις επιβολής όπου έχουμε συμφωνήσει ότι χρειάζεται ένα συστημικό πλαίσιο συνεργασίας σε ό,τι αφορά τη διαμεσολάβηση πάλι εκεί είναι ατελέστο σύστημα συνεργασίας μεταξύ διοικητικών αρχών και παρακαλώ εδώ λάβετε υπόψη ότι μιλούμε για διαμεσολαβήσεις μεταξύ αρχών και όχι μεταξύ ατόμων ή εργοδοτών κλπ. Το τρέχον σύστημα βασίζεται στο σύστημα διαμεσολάβησης κοινωνικών συστημάτων, όχι όμως για παράδειγμα στην απόσπαση. Και τέλος έχουμε κατακερματισμένο πλαίσιο συνεργασίας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε δηλαδή πολλούς επιμέρους μηχανισμούς, οργανισμούς, δίκτυα που συνεργάζονται αλλά όχι συστηματικά. Και εμείς μπορούμε να προσφέρουμε μια πιο συστηματική πλατφόρμα για μια πιο διαρκή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών που επιλαμβάνονται των διαφόρων τομέων. Έτσι, ο στόχος τώρα είναι να ενισχυθεί η δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη, αλλά πιο συγκεκριμένα να βελτιωθεί η συνεργασία, να ενισχυθεί η συνεργασία, η επιχειρησιακή συνεργασία, να προσφερθούν διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση στρεβλώσεων της αγοράς εργασίας, να καλύψουμε δηλαδή τα κενά τα οποία ανέφερα προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια για την αξιολόγηση, καλύτερου τρόπου δράσεως. Έχουμε βέβαια την αποτελεσματικότητα, έχουμε όμως και τα βασικά της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλαμβάνει μόνο την κατάλληλη και επαρκή δράση, χωρίς να οικειοποιείται αρμοδιότητες που είναι καλύτερο να παραμείνουν στο εθνικό επίπεδο. Και να πράξει μόνο τα αναγκαία. Αυτά είναι σημαντικά ω στοιχεία για την εκτέλεση των καθηκόντων. Έχουμε χωρίσει τη μελέτη δικτύπου σε δύο μέρη. Αφενός τα καθήκοντα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και το δεύτερο μέρος το πώς θέλουμε να εκτελεστούν τα καθήκοντα αυτά. Έρχομαι τώρα στα καθήκοντα. Νομίζω ότι αυτά τα εξήγησε ούτως ή άλλως η κυρία Τάισεν. Εδώ έχουμε χωρίσει κατά βάση σε τρία μεγάλα τμήματα επιλογών. Μπορείτε να πάρετε μια πιο light προσέγγιση, πιο ήπια, με κάποιες ελάχιστες ρυθμίσεις σε όλο το φάσμα των εγκαθηκόντων. Μπορείτε να προσαρμόσετε ενδεχομένω κάποια επιχειρησιακή ικανότητα και να διασφαλίσετε ότι θα καλυφθούν τα κενά με δράσεις που μπορούν να αναλαμβάνονται ακριβώς για να καλυφθούν τα κενά αυτά με πιο συγκεκριμένο και κατάλληλο τρόπο και τέλος υπάρχει και η επιλογή της εποπτείας που σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες αρχές εποπτείας επί των χωρών μελών πέραν των όσων προβλέπονται τώρα στο εφιστάμενο πλαίσιο. Δεν θα εξηγήσω τις επιπτώσεις σε προϋπολογισμό και σε στελεχικό δυναμικό. Βλέπετε ωστόσο τα νούμερα. Θα χρειαστεί κάποια επιβάρυνση του προϋπολογισμού γιατί στείλουμε ένα καινούριο σύστημα. Η τρίτη επιλογή είναι και η πιο δαπανηρή διότι απαιτεί ένα αριθμό δράσεων από πλευρά τη Επιτροπή. Γιατί ζητούμε λοιπόν, γιατί προτείνουμε καλύτερα την επιχειρησιακή επιλογή, διότι είναι ένας ε, ορθός συμβιβασμό ανάμεσα στις φιλοδοξίες και στο κόστος. Είναι αναλογική και όπως είπαμε αυτό είναι κριτήριο κλειδί για την επιλογή η επιλογή που επιλέγουμε, α το πούμε έτσι, είναι ε, καλύτερη από την πρώτη και λιγότερο δαπανηρή από την τρίτη. Αν προχωρήσουμε τώρα στην υλοποίηση, μιλήσαμε για τρεις δυνατότητες βασικά. Μία μπορεί να είναι να μην γίνει καθόλου οργανισμός. Να προχωρήσουμε απλώς σε βελτίωση της ε, συνεργασίας μεταξύ των υφισταμένων δικτύων και να δοθεί ένας βελτιωμένο ρόλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων. Μπορεί κανείς μετά να ιδρύσει αρχή, οργανισμό, όπως θέλετε πέστε το, με επιχειρησιακή δράση και μπορεί κανείς τέλος να δημιουργήσει την αρχή αυτή βασισμένη στις υφιστάμενους οργανισμούς, στις υφιστάμενες αρχές εργασίας. Συζητήσαμε τις τρεις αυτές επιλογές Αυτές βέβαια έχουν και διαφορετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ασφαλώς φτιάχνουν ένα δίκτυο που συναπαρτίζεται από τα διαφορά άλλα δίκτυα είναι και η λιγότερο δαπανηρή επιλογή, διότι δεν συμβαίνει ότι στείνεται από την αρχή ένα καινούριο σύστημα. Βέβαια θα χρειαστεί περισσότερο προσωπικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειάζονται περισσότεροι πόροι, δηλαδή δεν είναι εντελώς ουδέτερο δημοσιονομικά. Και τονίζω επίσης ότι η δημιουργία, επιλογή τρία τώρα, της δημιουργίας της αρχής πάνω σε μια εφιστάμενη αρχή οργανισμό, δεν θα είναι και πολύ λιγότερο δαπανηρό από το να φτιαχτεί μια αρχή από την αρχή, δηλαδή εξ αρχής με την έννοια αυτή, γιατί έχουν τελείως διαφορετικό στόχο και διαφορετικά καθήκοντα. Δηλαδή θα πρέπει να φτιάξει κανείς νέα καθήκοντα και να προσλάβει νέο προσωπικό πέραν των υφιστάμενων οργανισμών ή αρχών. Η επιλογή λοιπόν που επιλέγουμε τελικά είναι να δημιουργηθεί μια νέα αρχή που είναι και πιο ισορροπημένη και από την άποψη του κόστους. Προβλέπουμε ένα προσωπικό της τάξης των 144 προσώπων που βλέπετε ότι σε σύγκριση με άλλους οργανισμούς είναι μεν παραπάνω από τους άλλους οργανισμούς που ασχολούνται με την απασχόληση, είναι όμως και πολύ λιγότερο αριθμητικά από άλλους οργανισμούς, ο Frontex για παράδειγμα, η Eurojust. Ο προϋπολογισμός επίσης είναι ασφαλώς πολύ πιο περιορισμένος, πολύ μάλλον σημαντικότερο σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς απασχόλησης, αλλά πολύ μικρότερο από τον Frontex, για παράδειγμα, που έχει επιχειρησιακές δραστηριότητες πολύ σημαντικές. Θέλω μόνο να αναφέρω ως ε, τελική παρατήρηση ότι άνω του 50% του προϋπολογισμού που προβλέπεται για την ELA θα κατευθύνεται σε επιχειρησιακό κόστος, ενώ οι άλλοι μηχανισμοί, βασικά οι άλλοι οργανισμοί, κυρίως δαπανούν τα χρήματα που λαμβάνουν για δαπάνες προσωπικού. Και εδώ βεβαίως υπάρχει ένα τμήμα σημαντικό δαπανών προσωπικού, αλλά δεν είναι το κύριο. Διότι θα δίνεται κυρίως για διεξαγωγή επιθεωρήσεων, όπου κάνατε και πολλές ε, ερωτήσεις στην κυρία Τάισιν σχετικά. Αυτά από μένα για την ώρα και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Πανκάλντη της Γενικής Διευθύνσεως για την απασχόληση. Θα δώσω το λόγο για σύντομη παρέμβαση στην κυρία Λεξία Μανιάκη Γρίβα. από την, ε, την υπηρεσία του Κοινοβουλίου, την υπηρεσία έρευνας του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που μας καλείτε να παρουσιάσουμε την αρχική μας εκτίμηση για την αξιολόγηση αντιχτύπου. Πριν παρουσιάσω τα βασικά σημεία της αξιολόγησής μας, ακροθυγώ να επενθυμίσω ποια είναι αυτή η αρχική εκτίμηση και πώς ε, στηρίζει η μονάδα μας τα μέλη. Λοιπόν, δίνουμε αρχικές εκτιμήσεις αξιολογήσεως εκτι... ε, συνεπιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολογούμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, τα ισχυρά και αδύναμα σημεία, να αξιολογήσουμε την ποιότητα της αξιολογήσεως αντιχτύπου και κατά πόσο συνάδει με τους κανόνες και κριτήρια την αξιολόγηση αντιχτύπου καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για καλύτερη νομοθεσία. Δεν αξιολογούμε την ουσία της προτάσεως αυτή καθ' αρχική εκτίμησή μας στόχο έχει να δώσει ε, ανάλυση κατά πόσο η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα στοιχεία που παρέχω τη αξιολόγηση αντικτύπου είναι ορθά στοιχεία και χρήσιμα για την ε, εξέταση τη προτάσεω, αλλά δεν συζητούμε θέματα διαμορφώ πολιτική αρχαία αξιολογήσει. Είναι προ ενημέρωση και για υπόβαθρο για να βοηθήσουμε τι κοινοβουλευτικέ επιτροπέ και τα μέλη του Κοινοβουλίου στο έργο του. Πέραν αυτού, πέραν αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση κατόπιν ετήματος των μελών και αποφάσεως των συντονιστών η μονάδα παρέχει και, προς, και συμπροματική αξιολόγηση υποκατάστατο της των συνεπειών και των συνεπειών που έχουν τροπολογήσει του Κοινοβουλίου. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα, στην αξιολόγηση συνεπειών για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασίας, ξεκινώντας από τα βασικά στοιχεία. Οποιαδήποτε αξιολόγηση αντιχτύπου έχει σημαντικότητα τη συνιστόσα. Ορισμός του προβλήματος είναι αυτό. Σχετικά με αυτό, πιστεύουμε εν γέννη ότι η αξιολόγηση αντιχτύπου παρουσιάζει λογικά την προσέγγιση όσον αφορά την πρωτοβουλία και τα προβλήματα που θα λύσει η δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ο συνάδελφο ανέφερε ήδη τα προβλήματα. Ανεπαρκή πληροφόρηση, προσανατολισμό, στήριξη, προβλήματα συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών σε διασυνοριακέ περιπτώσει. Ο ορισμό του προβλήματο είναι καλά τεκμηριωμένο, υποστηρίζεται από διάφορε εκθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπέ, μελέτε, στατιστικά στοιχεία, και αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους κύκλους. Η εξολόγηση συνεπιών συμπεριλαμβάνει πολύ χρήσιμη ανάλυση και σχετικό έγγραφο στο παράτημα 12. Εκεί παρουσιάζονται πρόσφατα στοιχεία για την κοινικότητα του εργατικού δυναμικού και εξηγούνται δυσκολίες οι και το μέγεθος ε, της αδήλωσης εργασίας και της απάτης. Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει με χρήσιμο τρόπο τα προβλήματα και την κλίμακα των ε, προβλημάτων οι έξι συνιστώ των προβλημάτων καθορίζονται, αλλά περαιτέρω διευκρινήσεις θα χρειαζόταν σχετικά με το πρώτο πρόβλημα, ανεπαρκού ενημέρωση και προσανατολισμού. Κατά την άποψή μα, η αξιολόγηση συνεπιών δεν εξηγεί επακριβώς επακριβώ που χρειαζονται πληροφορίε που κενά και κατά συνέπεια δεν παρέχονται επαρκή στοιχεία στην κλίμακα των προβλημάτων και άλλες εξηγήσει και παρουσίασης πληροφοριών και δυσκολιών και κενών στις δράσεις τα εφιστάμενα εργαλεία θα ήταν κάτι ευπρόσδεκτο διότι υπάρχουν ήδη αρκετά διαθέσιμα εργαλεία και άλλα εργαλεία που επίκενται όπως η ενιαία πύλη για τα ψηφιακά ή το σχέδιο δράση Solvit. Εν γέννη, κατά την άποψή μας, το δεύτερο εντοπιστό πρόβλημα για τη συνεργασία μεταξύ αρχών. Τα προβλήματα συνεργασία αρχών είναι πιο καλά τεκμηριωμένα τα προβλήματα αυτά από ότι το προηγούμενο. Τώρα η δικαιολόγηση για τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ενώση και προ τη είναι αξία. Και τα θέματα επικουρικότητα και αναλογικότητα. Αυτά τα θέματα παρουσιάζονται στην εξολόγηση αντικτύπου σε συγκεκριμένο τμήμα. Έτσι θα έπρεπε, σύμφωνα στου αντολισμού, παρόλο που το τμήμα αυτό είναι αρκετά Βραχή όσον αφορά την αναλογικότητα αυτή η πτυχή ελήφθη υπόψη στη συζήτηση των διαφόρων επιλογών πολιτικής και ήταν στους παράγοντες που οδήγησε στην επιλογή της ε, ε, προσέγγισης που τελικά προτιμήθηκε. Όσον αφορά τους στόχους της επιλογές, εξολόγηση συνεπιών καθορίζει γενικού στόχου επιχειρησιακού και συγκεκριμένου σύμφωνα με του προσανατολισμού για καλύτερη νομοθεσία. Επιχειρησιακοί στόχοι που συνδέονται με του με τα προτινόμενα καθήκοντα τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασία βρίσκεται στο τμήμα τη αξιολόγηση με διάφορου σχετικού δείκτε. Κατά την άποψή μα, οι στόχοι έχουν σαφή σχέση με τα καθοριστέντα προβλήματα. Τώρα, όσον αφορά τι επιλογέ που συζητήθηκαν για την επίτευξη των στόχων, έχουμε δύο ομάδε επιλογών που συζητούνται. Από την πλευρά, επιλογέ όσον αφορά τα καθήκοντα πρέπει να εκτελεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εργασία και επιλογέ όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η εν λόγω αρχή. Σε κάθε περίπτωση η αξιολόγηση συνεπιών αξιολογεί τρεις επιλογές, πέραν της καθιστική τάξης και κατά άποψή μα επαρκεί ένα ευρύ φάσμα ε, επιλογών. Αυτές οι επιλογές απορρέουν από τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένου κύκλου και συνδέονται σαφώ με του στόχου και τα προβλήματα προ επίλυση. Όμως, Φρονούμε ότι οι περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές και συγκεκριμένα όσον αφορά τις επιχειρησιακές πτυχές των καθηκόντων της αρχής θα ήταν κάτι πρόσδεκτο. Πιο συγκεκριμένα, ε, εκεί που αναφέρεται η επιλογή 2 για την επιτέξη των στόχων, δηλαδή η δημιουργία νέας υπηρεσίας βάσει φυσταμένων δομών, η αξιολόγηση συνεπιών παρέχει περιγραφή του ρόλου της αρχής και προσπαθεί να εξηγήσει πώς οι δραστηριότητε αυτές θα συμπεριληφθούν σε άλλε πολιτικέ θα συντονιστούν. Κατά την άποψή μα όμω, λεπτομερέστερη διευκρίνηση και πιο συγκεκριμένη διευκρίνηση θα ήταν χρήσιμη όσον αφορά το ρόλο τη αρχή σε συνάρτηση με διάφορε άλλε υφιστάμενε δομέ και εργαλεία. Διότι πολλοί εμπλεκόμενοι φορεί εξέφασαν ανησυχίε για ενδεχόμενου κίνδυνου αλληλεπικάλυψη και ε, περιπλοκότητα διοικητική. Η επιλογή 3 θα δημιουργούσε την αρχή μέσω συγχωνεύσεως της με υφιστάμενο φορέας στον τομέα της πολιτικής ε, απασχόλησης. Η εν λόγω επιλογή ε, εξηγείται στην αξιολόγηση και γιατί δεν επιλέγεται αυτή η επιλογή. Αναφέρει η αξιολόγηση αντικτύπου ότι οι φυστάμενοι ε, φορείς δεν έχουν διασυνοριακή εξειδίκευση και βασίζονται στην έρευνα και αποτελούνται από τρία τμήματα και αυτό δίνει ιδεώδης δομή για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης, εργασία συγγνώμη. Και θεωρεί δυσανάλογη την αναδόμηση των φορέων μόνο για να επιληθούν προβλήματα σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων. Όμως αργότερα αναφέρει ότι η προτίμηση για την επιλογή 2, δηλαδή νέα υπηρεσία, δεν αποκλείει μελλοντικέ αποφάσει να δημιουργηθεί μια νέα αρχή βάση υφιστάμενου αποκεντρωμένου φορέα. Η εξολόγηση ποιόν εξηγεί ότι με τέτοια απόφαση θα έπρεπε να συμπληρώνεται μετά την συμπλήρωση εξολόγηση των υφισταμένων αποκεντρωμένων φορέων στον τομέα τη απασχόληση. Αυτό μα κάνει να διαρωτώμεθα. Μήπω θα ήταν καλύτερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμένει για, περιμένει για τα αποτελέσματα τη λόγω αξιολογήσεω που τώρα έχει ολοκληρωθεί πριν προτείνει το παρόν, την παρούσα λύση. Εν γέννη, περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις πτυχές ε, θα ήταν ενδιαφέρουσες. Τώρα σχετικά με τον αντίκτυπο που αξιολογείται. Όλες οι επιλογές αξιολογούνται οικονομικά, δημοσιονομικά, κοινωνικά και νομικά καθώς και όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως την προστασία των δεδομένων συγκρίνονται έναντι των κριτηρίων για αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και συνοχή σύμφωνα με τι κατευθυντήρε γραμμέ για καλύτερη νομοθεσία. οικονομικό αντίκτυπο γίνεται για του εργοδότε, μικρομεσαίες επιχειρήσει και εθνικού φορεί, Σύμφωνα με την αξιολόγηση συνεπιών, οι εταιρείε και κυρίω μικρομεσαίες επιχειρήσει ωφελούνται από πιο θεμητό ανταγωνισμό και από ισότιμου όρου και για από τη μείωση τη αβεβαιότητα σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων. Οι δημοσιονομικέ συνέπειε επεξηγούνται διαφανώ και αναφέρονται και υπολογισμοί και υποθέσεις. Ο προπολογισμό που υπολογίζεται είναι η μόνη ποσοτικοποιημένη αξιολόγηση. Υπάρχουν κάποιες διαφορές μεταξύ του ποσού που αναφέρεται στη σύνοψη, στο επόμενο μας προτάσεως και αυτού που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της αξιολογής συνεπειών. Εκεί αναφέρεται ότι το τίσιο ποσό, το τίσιο κόστος είναι περίπου 54 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η πρόταση αναφέρεται στα 50,9 εκατομμύρια. Τώρα, η ποιότητα των στοιχείων στην αξιολόγηση ποιον και η ποιότητα της αναλύσεως αυτή, αυτής καθ' εξηγείται η τεχνογνωσία που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι χρησιμοποιεί εσωτερικό αναλυτικό δυναμικό και φυστάμενες συμβάσεις. Οι μελέτες που χρησιμοποιήθηκαν ε, αναφέρονται αλλά δεν δίνονται διασυνδέσεις ε, στο διαδίκτυο και γίνεται πιο περίπλοκη έρευνα. Θεωρούμε τα στοιχεία που παράσχονται είναι νοπά ε, και είναι σωστή πηγή ενημέρωσης. Η εξολόγηση αντικτύπου ακολουθεί ποιοτική προσέγγιση και είναι διαφανή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξηγεί διότι σχέση και και αιτιατού για την υπηρεσία δεν είναι κάτι σαφές, δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Δεν αναφέρονται οι οικονομίες που θα απέρευσαν από απλούστευση και από τη βελτίωση αποδοτικότητας και εξηγεί έκθεση ότι δεν έκανε αυτό για λόγους ε, χρονικού περιορισμού, χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες όμως, στην αλλάση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. <coughs> Σχετικά με τη διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους κύκλους δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε προσπάθειες για διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους κύκλους, το βαθμό του δυνατού. Ήταν ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση. Διερευνήθηκαν οι απόψει των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία τη εν λόγω υπηρεσία εργασία. Αυτή η διαβούλευση όμω διήρκεσε μόλι 6 εβδομάδε, αντί 12 εβδομάδε που απαιτούνται κανονικά από τι κατευθυντήριε γραμμέ για καλύτερη νομοθεσία. Πέραν αυτού, στοχευμένη διαβούλευση έγινε διαβούλευση με αυτούς που εφαρμόζουν τα μέτα, δημόσιες αρχές, πολίτες, κοινωνικούς εταίρους και άλλη διαβούλευση έγινε συγκεκριμένα για τον τομέα των μεταφορών. Αυτό αφορούσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι οι περισσότεροι εμπορευόμενοι στον τομέα των οδικών μεταφορών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά τι στοχευμένε αυτές διαβουλεύσεις, θα ήταν χρήσιμε περισσότερες πληροφορίες για εκείνους που έδιναν, έδιναν τις αριθμό απαντήσεων, αυτά λείπουν στην αξιολόγηση. Επίσης, οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν τοποθετήθηκαν για επιλογές γρήγορων ταχαίων αποτελεσμάτων, τι μορφή θα έπρεπε να έχει αυτή η αρχή, αλλά εξέφρασαν όμως οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι μικτές απόψεις σχετικά με τις οργανωτικές πτυχές της εν λόγω αρχής. Εν γέννη, οι απόψει των εμπλεκομένων φορέων αναφέρονται σαφώ στου ανάλογου τομεί για τι επιλογέ και τον καθορισμό των προβλημάτων, καμιά φορά πολύ γενικόλογα, με φράσεις όπως σημαντικός αριθμός εμπλεκομένων ή πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς χωρίς να αναφέρονται συγκεκριμένοι αριθμοί και κατανομή των αριθμών αυτών. Κλείνοντας, θεωρούμε ότι η πολυ εμπλεκομενοι φορεις χωρις να αναφερονται συνεπιών ε, παρουσιάζει λογικά την πρωτοβουλία, τη λογική που ακολουθήθηκε και τη δράση που επιβάλλεται από πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Καθορίζονται μέσω στοιχείων τα προβλήματα, μέσω μελετών, μέσω διαβουλεύσεων με του εμπλεκομένου φορεί χρειαζόνται περισσότερα στοιχεία για τι ανάγκε και τυχόν κενά. Εξολόγηση συνεπιών καθορίζει σωστά τα προβλήματα, δικαιολογεί την παρέμβαση, καθορίζει του στόχου και τι επιλογέ. Όλα αυτά τα κάνει σωστά και τεκμηριωμένα. Λεπτομερέστερη περιγραφή όμως των επιλογών και επιχειρησιακών πτυχών θα ήταν κάτι επωφελές για την ανάλυση εξολόγηση αυτή των συνεπειών θα έπρεπε να εξηγήσει καλύτερα γιατί θεωρεί ότι θα ήταν δυσανάλογο να αναθεωρηθούν οι φορεί μόνο για την επίλυση προβλημάτων για την κινητικότητα των εργαζομένων και μετά θεωρεί όμω ότι η προτίμηση τη επιλογή 2 δεν αποκλείει μελλοντικέ αποφάσει να δημιουργηθεί νέα αρχή επιφυσταμένων αποκεντρωμένων φορέων, κάτι που συζητείται στα πλαίσια τη επιλογή 3. Εξολόγηση αντιχτύπου, ακολούθησε τι συστάσει για βελτιώσει που ζήτησε ρυθμιστικό φορέα θα έπρεπε να συζητήσει περισσότερο τον κίνδυνο περιπροκότητας και επικάλυψης καθώς και ενδεχόμενη συμπερίληψη αυτών των τυχών και συνεργειών των διαφόρων φορέων ε, που υπάρχουν με την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι καλύτερες πληροφορίες, πιστεύουμε. Τέλος, εξολόγηση αντικτύπου δείχνει ότι οι προσπάθειες κατεβλήθησαν για την άποψη των εμπλεκομένων φορέων, παρόλο που η διαβούλευση δεν διήρκεσε όσο θα έπρεπε 12 εβδομάδε και απόψη των μπλεκομένων φορέων εν γέννη αντικατοπτρίζονται καλά στο κείμενο όσα αναφέραν προηγουμένως αυτά τα πορίσματα αφορούν μόνο τα ισχυρά και ασθενή σημεία της εκθέσεως αξιολογήσεως αντιχτύπου και ουχή την ουσία της προτάσεως. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ε, Mr. Ευχαριστώ. Κύριε Λέναρς, θέλετε να κάνετε καμιά ερώτηση. Uh, Ευχαριστώ πολύ και για τις δύο παρουσιάσεις. Ε, ενδιαφέρουσα επιλογή ανάμεσα στη δεύτερη εκδοχή και στην τρίτη. Operational και supervisional, δηλαδή επιχειρησιακή λειτουργία η εποπτική. Μπορεί να, υπάρξει κάποια, να έχει υπάρξει κάποια παρεξήγηση, παρανόηση για τις πραγματικές εξουσίες και το ρόλο αυτής της αρχής. Το είδαμε και από τη συζήτηση με την κυρία Τάισεν και το πρόβλημα είναι από την ονοματολογία. Όταν ονομάζεις κάτι authority, αρχή, αυτό σημαίνει ότι έχει την αρχή και το κύρος και την εξουσία να ε, παίρνει κάποιες αποφάσεις, να τις επιβάλλει και στη συνέχεια να προβαίνει σε κυρώσεις. Και αυτά τα περί κύρους και αρχής μου θυμίζουν και τη μητέρα μου. Γιατί αποφασίσατε να το βαφτίσετε authority, ενώ δεν είναι αρχή με την έννοια που αντιλαμβανόμαστε ή στην πρόταση όπως έχει υποβληθεί. Ε, και σε ό,τι αφορά την παροχή ε, πληροφοριών και ενημέρωσης, είναι ενδιαφέρον ε, κάποιο που θέλει να περάσει σύνορα για να ε, εργαστεί να έχει τη σωστή ενημέρωση και την αναγκαία. Αλλά αυτό πραγματικά πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ τη μελέτη αντικτύπου, αν χρειάζεται να ενημερώνεται ο πολίτης. Δεν μπορεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο ή σε εθνικό. Ρώτησα και την κυρία Επίτροπο προηγουμένω, την κυρία Τάισεν. Αυτά ρυθμίζονται από φορολογικέ, διμερεί φορολογικέ συμφωνίε μεταξύ κρατών μελών. Έχω μια ερώτηση για το άρθρο 14, συνεργασία σε περίπτωση ε, διατάραξης της αγοράς σε διασυνοριακές ε, περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Και μετά τη μελέτη αντικτύπου, για ποιο λόγο βάλετε τέτοια διάταξη στο κείμενο. Έτσι, μερικές μόνο ερωτήσεις αυτές. Ευχαριστώ, μην ξεχνάτε ότι, ε, τις ερωτήσεις του κυρίου Λέναρς θα δώσω το λόγο και σε άλλους συναδέλφους και στον κύριο Πυρίνσκι. Ε, σημειώστε τις για να απαντήσετε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Η δική μου ερώτηση έχει σχέση ακριβώς με πώς, το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια της επιβολής ε, του νόμου που κρύβεται πίσω από την πρόταση. Η Επίτροπος Τάισεν εδώ, τις παρατηρήσεις προηγουμένως, ανέφερε δύο-τρεις φορές την έννοια της εμπιστοσύνης μεταξύ της αρχής αυτής και των εθνικών αρμοδίων αρχών. Και αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε όταν συζητούμε τις δομές και το ρόλο και τις αρμοδιότητες αυτού του οργανισμού να τα λάβουμε υπόψη. γιατί θυμάμαι από την εμπειρία που είχαμε με την πλατφόρμα για την άδειλη εργασία, την ότι έλεγαν ορισμένοι ότι δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Γιατί αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα. Μετά καταφέραμε όμως να επιχειρηματολογήσουμε και να πούμε ότι εδώ έχουμε σύμπτωση συμφερόντων εργαζομένων εργοδοτών και κρατικών αρχών. Του συμφέρει όλους να τηρούν ε, με απλό τρόπο και αποτελεσματικό τους κανόνες. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στη δεύτερη από τις τρεις επιλογές για το ε, ε, ρόλο και τη φύση του οργανισμού. Και μία αρχή θα πρέπει να έχει ακριβώς το κύρος που μπορεί από το ρόλο της και να ε, δημιουργεί εμπιστοσύνη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω τώρα, αλλά αυτό θα πρέπει να φαίνεται παντού. Έχει να κάνει και με την Επιτροπή Ενδιαφερομένων Κύκλων. Ε, από τη δημιουργία της αρχής να δούμε πώς θα γίνεται η μεσολάβηση. Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Γιατί έχουμε μόνο έναν εκπρόσωπο των κρατών μελών και δύο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ποιο λόγο περιορίζονται τα κράτη-μέλη με συγκεκριμένες προϋποθέσεις για το ποιους υπαλλήλους ε, μπορούν να αποσπάσουν, ενώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Ποιος θα ορίσει τον εκτελεστικό διευθυντή, ε, μετά από πρόταση μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί μόνο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυβερνήσεις. Στην ομάδα εκεί των ενδιαφερομένων κύκλων. Ε, είναι και οι κοινωνικοί εταίροι εκεί που εκπροσωπούνται. Ναι, αλλά με, με βάση την τριμερή εκπροσώπηση. Δηλαδή, κυβερνήσει, εργοδότε, εργαζόμενοι. και αυτά ποιος θα τα φροντίζει και ποιος θα τα ορίζει ο, ο εκπρόσωπος ή ο πρόεδρος στην διαχειριστική επιτροπή ή κάποιος από το Συμβούλιο. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα που θέλω να ρωτήσω για να διευκρινίσω. Δεύτερον, ωραία εμπιστοσύνη και καλή, αλλά θέλει και λίγο βούρδουλα. Υπάρχουν πολύ ευαίσθητοι τομεί, α πούμε, σαν γι' αυτό. Δεν αρκεί εμπιστοσύνη. Θέλει και ένα φόβητρο. Έχετε σκεφτεί να εμπνευστείτε από άλλες εποπτικές αρχές, ας πούμε στην προστασία των καταναλωτών. όπου υπάρχει πολύ περιγεγραμμένη διατύπωση ε, σωστά δηλαδή και με ουσία για το τι ρόλο έχουν τα ευρωπαϊκά όργανα, τα εποπτικά και πώς θα ενισχυθούν οι εθνικές αρχές στη συνέχεια. Διότι ξέρουμε ότι με την κρίση και όλη αυτή τη λιτότητα που ζήσαμε είναι υποστελεχωμένα και υποχρηματοδοτούμενα αυτά τα όργανα και νομοθετικά πιο αποδυναμωμένα δεν θα μπορούσε η αρχή να κοιτάξει λίγο τι γίνεται με τη δυνατότητα της εκάστοτε διοικητικής κρατικής μηχανής να αντιδράσει, γιατί έχουν διαφορές από χώρα σε χώρα. Θα πρέπει να ευαισθητοποιεί, να ενθαρρύνει ε, τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων δομών στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακλάται και ε, στις συστάσεις αναχώρα για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Και να δούμε φυσικά επίσης και όλο το φάσμα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και ποια είναι αυτά τα άρθρα στη ΣΛΕ, τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω το 81 και το 82 είναι. Το αναφέρει ένα από τα έγγραφα για την ενισχυμένη επιβολή και την δικαστική συνεργασία σε θέματα αστικού αλλά και ποινικού δικαίου. Και καλό είναι να ασχολείται με το ποινικό σκέλος, γιατί ένα πρόβλημα από την αδήλωτη εργασία εμπίπτει στο κοινό ποινικό δίκαιο. Kind of So the, the by in... Και η αρχή θα πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά και θα μπορούσε να, να ενισχύσει αυτή η αρχή την ίδια της στην αρχή και το κύρος. Και το σημείο 3, Πρόεδρε, έχει να κάνει με το εξή για την λεγόμενη αυτή συμβουλευτική ομάδα επιτροπή. Τι είναι αυτό το πράγμα, θα μπορούσατε να επεκταθείτε λίγο, διότι μαθαίνω εδώ από δεξιά και αριστερά ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να εμπλακεί στη νομοθετική διαδικασία για τον προτινόμενο κανονισμό. Στόχο έχει να εξασφαλίσει και να βεβαιωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση που και όταν εγκριθεί ο κανονισμός. Όλα αυτά είναι ε, πολύ ωραία και αξιοθαύμαστα, αλλά τι εννοείται ακριβώς. Ευχαριστώ. κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την παρουσίαση αυτή. Θέλω να επανέλθω λίγο στο θέμα της ενημέρωσης και τη συνεργασία ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο IMI και το ESSI. Αυτά είναι τα συστήματα που θα συντονιστούν. Παράδειγμα, αν δούμε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, αυτή από μόνη της θα ήταν ένα είδος ταυτότητας ευρωπαϊκής, οποιασδήποτε μορφής. Αλλά έτσι όπως έχουν τώρα τα πράγματα στο IMI, το ESSI και τις καθυστερήσεις και όχι μόνο καθυστερήσει και παραπάνω στην κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Θεωρείτε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τα εφιστάμενα συστήματα και τις ατελείς πληροφορίες που έχει. Ε, άκουσα τι είπε η Υπηρεσία Ερευνών του Κοινοβουλίου λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκτιμήσει σωστά τα ε, ελλείμματα ε, στην κλίμακα αυτή της πληροφόρησης. Ξέρουμε ότι υπάρχει ε, έλλειμμα πληροφόρησης, αλλά δεν ξέρουμε τι τάξη μεγέθους είναι αυτή. Και όπως σας είπα, τα συστήματα είναι κατακαιρματισμένα και ατελή. Και με ενδιαφέρει αυτό και με ανησυχεί. Όταν χρησιμοποιείται έννοιες όπως αποτελεσματική και αποδοτική για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, Καλά θα κάναμε να αφιερώσουμε περισσότερες προσπάθειες στον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει σωστά από την αρχή αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω αν έχετε σχόλια από αυτού. Δεύτερον, και πάλι, ο συνάδελφος από το Κέντρο Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας είπε για την ε, αξιολόγηση των αποκεντρωμένων οργανισμών, η οποία ε, διατίθεται. Δεν την έχω δει. Κατά την άποψή σας, υπάρχει τίποτα στην αξιολόγηση αυτή που να μπορεί να βελτιώσει την πρόταση ως έχει. Και τρίτον, μιλήσατε για το λόγο των ε, λειτουργικών δαπανών προς τις ε, ουσιαστικές. είπατε ότι θα είναι περισσότερο από το μισό. Ε, πόσο περισσότερο. Και για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που θα τις κάνει. Ωραία όλα αυτά που μας λέτε, αλλά οι άνθρωποι είναι κάποια πρόσωπα αυτοί οι επιθεωρητές, οι ελεγκτές. Και αν δείτε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, όπου μιλούμε για συνεργασία, για διαμεσολάβηση, για δημιουργία ικανοτήτων, όλα αυτά είναι αποστολές με πάρα πολύ μεγάλη ένταση εργασίας. Επίσης αναλαμβάνει να διαχειριστεί κάποιες άλλες δομές που υπάρχουν και οργανισμούς, όπως είναι το EURES. Και λέτε ότι οι λειτουργικές δαπάνες, ε, ε, μάλλον το κόστος του προσωπικού θα είναι λιγότερο από το μισό του συνολικού. Αυτό λίγο με προβληματίζει, γιατί θα έχει πάρα πολλή δουλειά. Ε, προσωπικό θα έχει. και μια που μιλάμε για υπαλλήλους και προσωπικό. Ποιους θα επιβλέπουν, ποιους θα εξετάζουν τους. Στις 9 Φεβρουαρίου ε, η Συμβουλευτική Επιτροπή έδωσε στην αρχή αρνητική γνωμοδότηση, ενώ στις 20 Φεβρουαρίου ήρθε να δώσει θετική. Την 21 εντάξει. Ε, πολύ κοντά χρονικά. Πώς έγινε αυτό. Τι αλλαγές έγιναν μέσα σε αυτές τις 10-11 μέρες για να ικανοποιηθεί ε, το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο για να δώσει το πράσινο φως. Η Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Να δώσω πάλι το λόγο στον κύριο Πανκάλντι που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ε, ετέθησαν περίπλοκες ερωτήσεις. Παρακαλώ ωστόσο να είστε σύντομος και σαφείς στις απαντήσεις σας διότι έχουμε βέβαια και ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο οφείλουμε να σεβαστούμε. Ορίστε παρακαλώ κύριε Πανκάντη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Πέρα από το όνομα, Τι εξουσίες έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να ασκήσει. Αρχή σημαίνει και κάποια ιεραρχία. Η ιεραρχία ωστόσο πρέπει να πλαισιώνεται μέσα στα πλαίσια δηλαδή των εξουσιών της Ένωσης. Ορισμένα καθήκοντα η Ένωση δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει για παράδειγμα επιθεωρήσεις έρευνες, να τα επιβάλλει στι χώρε μέλη και κτλ. Αυτό ανταποκρίνεται και στο κριτήριο τη αναλογικότητα, βέβαια που ισχύει για την πρότασή μα. Σε ό,τι αφορά τις πληροφορίε, έχουμε δύο διόδους μεταξύ επιχειρήσεων, προς επιχειρήσεις μάλλον και πολίτες και βεβαίως και μεταξύ αρχών των χωρών μελών. κατ' επανάληψη γίνεται μνήα στην μελέτη αντικτύπου. Αποφεύγουμε τις επικαλύψεις, αλλά πίσω από την εννέα πύλη υπάρχει μεγάλη δουλειά που γίνεται για να προσφέρεται επαρκές πλήθος πληροφοριών και η Επιτροπή σας έχει ασχοληθεί και με την απόσπαση εργαζομένων και γνωρίζει τη σημασία τη παροχή πληροφοριών και για την αρχική εφαρμογή αλλά και για την αναθεώρηση τη οδηγία. υπάρχει ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η ποιότητα της, των πληροφοριών προ πολίτε και εργοδότε είναι επαρκή σε όλε τι χώρε μέλη. Βεβαίω, οι χώρε μέλη είναι αρμόδιε να παρέχουν τι πληροφορίε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει στήριξη και να επιτρέπει την σύγκριση τη ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται από που παρέχονται από τι διάφορε χώρε μέλη. Ε, προς τους ε, πολίτες και εργοδότες. Σε ό,τι αφορά τους μηχανισμούς για την διοχέτευση των προφορίων μεταξύ αρχών, οι διάφοροι μηχανισμοί που υπάρχουν, είναι οι επιμέρους μεταβλητές. Υπάρχουν, λειτουργούν, βέβαια με κάποιες ελλείψεις, ο SSI ακόμα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά ο EMI γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις της πλατφόρμας της αδήλωτης εργασίας. Και χρειάζεται ενίσχυση του τμήματος αυτού για την αδήλωτη εργασία. Και εκεί θα κάνουμε την προσπάθεια να τα προωθήσουμε και να περιλάβουμε και τα διάφορα άλλα για τα εμπόδια. Η ιδέα είναι η Ευρωπαϊκή Αρχή θα υποστηρίζει τις εθνικές αρχές. Θυμίζω την υπόθεση Κατέρπιλα εδώ στο Βέλγιο πριν από λίγους μήνες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφερε υποστήριξη στις εθνικές αρχές και στις τοπικές αρχές για να δουν πώς μπορούν να αλλάξουν τη χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, να το κατευθύνουν σε κάποια συγκεκριμένη περιφέρεια ή πώ να ζητήσουν την, την ε, υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Τέτοια πράγματα μπορεί να κάνει για να υποστηρίξει και τι διάφορε τοπικέ και εθνικέ αρχέ, εκτό τώρα του ρόλου πολιτική Η απόφαση δηλαδή να διατεθούν κονδύλια είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμίου. Επίση Αυτά υποφύγεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα για την διακυβέρνηση, κύριε Πυρίνσκι. Ακολουθεί την κοινή προσέγγιση Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Αυτό είναι το βασικό. Η ομάδα ενδιαφερομένων μερών έχει συμβουλευτικό ρόλο όταν θα δημιουργηθεί η αρχή στην διαδικασία για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχουμε μια συμβουλευτική ομάδα η οποία ασχολείται ιδίω με τις δυσχέρειες της περιγραφής των οργανισμών και των καθηκόντων που θα αναλάβουν και το πώς θα συνεργαστούν αυτές, ε, αυτοί οι φορείς. Πρόκειται για τμήματα τα οποία δεν εντάσσονται στο νομοθετικό πλαίσιο. Αλλά προετοιμάζουν το έδαφος για τη λειτουργία του οργανισμού, της αρχής δηλαδή. Τέλος για το, για το δημοσιονομικό αντίκτυπο και το προσωπικό. Δύσκολη υπόθεση να κατανοήσει κανείς τι, ποια πράγματα θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή εργασία από αυτά που κάνουν τώρα οι κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, διμερεί συμφωνίε που υπάρχουν μεταξύ χωρών μελών, στις οποίες διμερεί συμφωνίες προβλέπονται και κοινέ επιθεωρήσει. Πόσε από αυτές τώρα θα αχθούν ώστε να, στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Αρχή εργασία, ώστε να τελούνται υπό την αιγίδα τη. Έχουμε βάλει το όριο και έχουμε πει αν έχουμε 100 κοινέ επιθεωρήσεις, ποιε θα είναι ένα χρόνο, πώς θα είναι ένα χρόνο, ποιο προσωπικό θα χρειάζεται, ποιοι πόροι χρειάζονται. Και από την βάση αυτή έχουμε καταλήξει σε ένα υπολογισμό και για τον προϋπολογισμό, μια εκτίμηση δηλαδή και του προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί και του προσωπικού. Και θα δούμε και στα επόμενα χρόνια αν χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό, λιγότερο, περισσότερο κονδύλια από τον προϋπολογισμό, λιγότερο. Θα πω μια τελευταία λέξη τώρα για τους οργανισμούς. Υπάρχει σημαντική διάθεση να διαχωριστούν οι συζητήσεις για να μην προκληθεί σύγχυση. Θέλουμε να ξεχωρίσουμε την συζήτηση περί ELA, να δούμε ακριβώς τι μπορεί να κάνει, ποια καθήκοντα μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας χωρίς να μπούμε στο ποια καθήκοντα θα λαμβάνουν άλλοι οργανισμοί. Βεβαίως αυτά τα πράγματα είναι ανοιχτά στο μέλλον για ε, μελέτη και ε, προβληματισμό. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα κυρία Γρήβα. Να απαντήσω στην ερώτηση κυρία Χάρκιν για την αξιολόγηση. Πρόσφατα ήταν διαθέσιμη, πολύ πρόσφατα μια, μόλις πριν από μια εβδομάδα διατέθη. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε το κείμενο ακόμα. Σχετικά με τα σχόλια του Συμβουλίου, πράγματι ήταν σύντομο ο χρόνος που πέρασαν τι γνωμοδοτήσεις, αλλά η μελέτη αντιχτύπου, όπως προβλέπετε, έχει ένα παράρτημα με πίνακα. Εκεί αναφέρεται πώς συμπεριέλαβε την άποψη του Συμβουλίου, του Διοικητικού και την αρνητική και τη θετική με επιφυλάξεις. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην αξιολόγηση αντικτύπου με συγκεκριμένη μνήμα των τμήματων των σχετικών που έγιναν οι τροποποίησεις για να ληφθούν υπόψη σχόλια. Κατά την άποψή μας, οι περισσότερες συστάσεις ελήφθησαν υπόψη. Όμως και άλλες πληροφορίες θα μπορούσαν να δοθούν κατά την άποψή μας όσον αφορά το θέμα της αλληλεπικάλυψης, ενδεχόμενης αλληλεπικάλυψης και δεχόμενων συνεργασιών με τους διάφορους υφιστάμενους φορείς και τη συμπερίληψη αυτών των πτυχών σε άλλες πολιτικές. Mm. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Όπως θα ξέρετε έχουμε πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα. Το απόγευμα σας ενημερώνω. Συνεδριάζουν σκιώδεις εισηγητές εξ όσων κατάλαβα και μαθαίνω στις 2 η ώρα και εμπειρογνώμονες που δεν μπόρεσαν ακόμα να πούν τίποτα. Είστε προσκεκλημένοι σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως και οι υπόλοιποι βουλευτές. Μπορείτε να πάτε να κάνετε ερωτήσεις και να συζητήσετε με τους ειδικού μας εμπειρογνώμονες. Ωραία. Θα σας δώσω τώρα από πέντε λεπτά στον καθένα για να μας κάνετε μια σύντομη εισαγωγή Και σας είπα μπορείτε να πάτε και εσείς στη συνεδρίαση των σκιωδών για να εμβαθύνετε και να ενημερώσετε σε μεγαλύτερο βάθος. Λοιπόν, ωραία, θα δώσω τώρα το λόγο στη Βανέσα Λάντεν. Να αρχίσουμε από τον κύριο Γιάνν Κρέμερς. Καλά από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου του Τίλμπουργκ. Θα μας μιλήσει για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και την επιβολή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, διότι τα έγγραφα είναι στη διάθεσή σας και σε έντυπη μορφή και στο διαδικτύο. Αυτό που θα ήθελα να κάνω είναι να σας δείξω μερικές διαφάνειες. Έχω ετοιμάσει πολλές, αλλά δεν θα τις δούμε όλες. Τι σημαίνει η πρόταση για τις ε, επιθεωρήσεις εργασίας και τους είδους τους επιθεωρητές εργασίας. Τι θα σημάνει ε, αυτό για τις κοινέ επιθεωρήσεις και την επιβολή του κοινοτικού κεκτημένου της αντίστοιχης νομοθεσίας. Αν δείτε τη μελέτη αντικτύπου θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποια ευρήματα που αναφέρονται εκεί σχετικά και είναι ευπρόσδεκτο το γεγονός ότι συνενώνονται διάφορα κατακαιρματισμένα μέτρα που υπάρχουν και ισχύουν που είναι έτσι σαν σιλό κάθετες δομές, ανεξάρτητες μεταξύ τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι συνενώνονται και σπάει ο κατακαιρματισμός και πολύ χρήσιμο. Ε, βασικός στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι, ή θα έπρεπε να ήταν πριν από 30 χρόνια ήδη, να εξασφαλίσουμε δίκαιη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όπως είπε και ο κύριος Γιούνκερ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε ε, τη δυνατότητα δράσης και τη νομική των αρμοδίων αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πολύ περιορισμένη φιλοδοξία. Και να δούμε τι συμβαίνει και αλλού στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτή τη στιγμή αποφασίσει μία αρχή ή ε, αποφανθεί ότι υπάρχουν παρατυπίες και γίνεται έρευνα στις αρμόδιες εθνικές αρχές τότε θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή εντολή, ευρωπαϊκή έγκριση για δράση, όπως συμβαίνει αλλού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό απουσιάζει τελείως από την πρόταση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν κοιτάξετε τις εμπειρίες με τις επιθεωρήσεις και τις κοινέ επιθεωρήσεις και τους ελέγχους αυτή τη στιγμή, οι αρμοδιότητες και εξουσίες των ελεκτών, των επιθεωρητών, είναι πάρα πολύ περιορισμένοι όταν θελήσουν να βγουν από την εθνική τους επικράτεια και να πάνε σε άλλη χώρα. Σε διάφορους τομείς. Όταν υπάρχουν κάποια κατασκευάσματα με ε, ε, εταιρείε γραμματοκιβώτια, μαϊμού κλπ, Στο Βέλγιο υπάρχει μία έννοια όταν θέλεις να πεις ότι κάποιος εμπέζει, η έκφραση είναι ότι παίζει με τα πόδια μου. Ε, ε παίζουν με τα πόδια τους. Ε, στα Ολλανδικά είναι αυτό. Ε, γιατί έρχονται και τους λένε ότι η εταιρεία μου εδρεύει σε άλλη φορολογική επικράτεια και δεν έχεις καμία δικαιοδοσία εδώ. Θα πρέπει λοιπόν να δίνεται η έγκριση ε, των αρμοδίων εθνικών αρχών που συνεργάζονται. Ένα δεύτερο είναι ότι δεν έχει εκπονηθεί καμία πολιτική επιβολής προστήμων και κυρώσεων. Ε, αν δείτε ποιου τομείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε, τι θέλουμε να πατάξουμε. Την κατάχρηση της ελευθερίας εγκατάστασης, την κατάχρηση της ελευθερίας παροχής υπηρεσιών, και την συνοριακή αντίστοιχη κινητικότητα των εργαζομένων. Μα αν δεν έχει πολιτική για την επιβολή προστήμων, καμία, η δική μου εμπειρία τι λέγει. Καλά, όταν υπάρχουν διοικητικέ κυρώσει, αυτέ πάνε ε, στον κάλαθο των αχρήστων ή στο γραμματοκιβώτιο του γραμματοκιβωτίου τη Μαϊμού εταιρεία. Και φυσικά δεν θέλουμε εμεί κάτι τέτοιο. Σταματώ εδώ για τελειώνει ο χρόνο μου. Τα υπόλοιπα θα τα βρείτε στο έγγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στη Βανέσα Λάντεν που εκπροσωπεί την εταιρεία ε, που αξιολογεί τις υπηρεσίες αυτές στα πλαίσια του Eures. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. I maybe first like to start Ας ξεκινήσω λοιπόν συνοψίζοντας τι είναι το EURES, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, δημιουργήθηκε το 1993. Στόχος η διευκόνιση της κινητικότητας στην Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας. Πώς, παρέχοντας πληροφορίες, συμβουλές, βοηθώντας ε, να ταιριάξουν οι ανάγκες εργοδοτών εργαζομένων. Είναι και μία πύλη το EURES στο διαδίκτυο. Περί αυτού πρόκειται μου ζητήθηκε να δω ποιος είναι ο αντίκτυπος για το Γιούρες από την ε, σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας. Οι προτινόμενες αλλαγές, για να το πω σύντομα, μέσω της δημιουργίας του ELA, για μας, έχουν τετραπλή συνέπεια. Βλέπουμε τη δημιουργία νέου σημείου διαπαφής, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συντονισμού που εδρεύει εντό Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μεταφερθεί πλήρω στο ELA και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού παρέχει υπηρεσίες οριζόντιες στήριξης στο EURES. Συντονίζει το έργο του EURES. Παρέχει κατάρτιση πληροφόρηση, ενημέρωση. Όλα αυτά θα μπουν στο ELA. Άλλη αλλαγή. Διαχωρισμός των ευθυνών όσον αφορά την πύλη, τη διαδικτυακή. Ό,τι σχετίζεται με το περιεχόμενο και το σχεδιασμό της πύλης θα μεταφερθεί στο ELA. Ό,τι σχετίζεται με τεχνικές λεπτομέρειες θα παραμείνει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα θα έχουμε ένα διαχωρισμό. Εποπτεία. Το ρόλο των παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Εξετάζουν τα θέματα της κινητικότητας των εργαζομένων. Τώρα αυτά θα εμπέσουν στην αρμοδιότητα της ELA. Εν συντομία τώρα να αναφερθώ στην προστιθέμενη αξία της προτάσεως για το EURES και κάποιες συστάσεις μετά. θέμενη αξία λοιπόν, όπως τα βλέπει τα πράγματα το Γιούρες. Μεγαλύτερη προσπάθεια κοινό στόχο. Επτά φορείς Ευρωπαϊκής Ενώσεως ενώνονται Άρα βέλτιστε πρακτικέ και ιδέε μπορεί να ανταλλάσσονται. Η υποστήριξη είναι πιο ολοκληρωμένη για τα κράτη-μέλη σε υπερεθνικό επίπεδο. Αποτελεσματικότητα. Θα υπάρχουν κέρδη. Θα μπορεί σαν μια θηρίδα να λειτουργεί το γιούρες για παροχή πληροφοριών και μέσω συνεργασίας και διαφόρων πρακτικών Μέσω κοινών προγραμμάτων θα βελτιωθεί η αποδοτικότητα. Θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιες δραστηριότητε οριζοντίου χαρακτήρα, υποστήριξης, που εφαρμόζουμε να βελτιωθούν. Λόγω συνεργασίας με άλλους φορείς. Κατάρτιση φερειπίν. Άλλη δυνατότητα οι περιορισμοί που έχει τώρα το Γιούρες, τα κενά στις θέσεις, η ε, αίτηση για κάλυψη θέσεων, η βιογραφικά κλπ. Ίσως εκεί βελτιωθεί η κατάσταση μέσω του νέου φορέα. Θα μπουν περισσότερες πληροφορίες στην πύλη αυτή τη διαδικτυακή περισσότερο θα ανήκουν σε επίπεδο κρατών μελών αυτές τις πληροφορίες, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη να δημοσιεύουν τα κενά, τις κενές θέσεις. Και θα κερδίσουμε σε αποδοτικότητα μέσω συνεργασιών που αναπτύσσονται επεκτείνοντας την πύλη του Γιούρες, κυρίως το τμήμα για συνθήκες διαβίωσης και εργασίας με τη συνεργασία των άλλων φορέων που θα εμπέσουν στα πλαίσια του νέου αυτού οργανισμού. Άλλα θετικά στοιχεία, η αξία, λόγω του ΙΑΛΕΗ. Θα δοθεί ευρωπαϊκό πρόσωπο στην ε, κινητικότητα των εργαζομένων. Θα προβληθεί το Γιούρες περισσότερο και τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόθεση της κινητικότητας των εργαζομένων πόρισμα της ECA, αλλά δεν ήταν τόσο όρατα αυτά τα στοιχεία όσο θα γίνουν τώρα. Σε μία για περαιτέρω προβληματισμό. Να δημιουργηθεί άλλο ένα σημείο διαπαφής. σχετικά με κάποιες αλληλεπικαλύψεις που υπάρχουν και την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού και διευκρινήσει των διαφόρων ρόλων. Σημαντικό. Κυρίως για το EURES και σε σχέση με το ENPS, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Υπηρεσιών για την Απασχόληση στο Δημόσιο Τομέα και ενδεχόμενη αλληλεπικάλυψη μεταξύ των ε, ε, διαφόρων εθνικών ε, φορέων συντονισμού και των εθνικών αξιωματικών συνδέσμων που θα ενταχθούν στη νέα υπηρεσία. Κάτι άλλο. Η οργάνωση, η επιμελητία όσον αφορά τη γεωγραφική κατανομή των ευθυνών. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Επιμερισμός των ευθυνών στην πύλη τη διαδικτυακή. Και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Και πώς θα γίνει ο χειρισμός αυτής της προσπάθειας. Σαφήνεια απαιτείται για τους πόρους, για το γιούρες. Θα αυξηθούν, θα ενισχυθούν οι πόροι. Οικονομική διαχείριση. Να αποφευχθεί αύξηση του διοικητικού άχθους για τα κράτη-μέλη. Οι συστάσεις που έχουμε απορρέουν από όλα αυτά τα σημεία που σας παρουσίασα και αναφέρονται στο ενημερωτικό έντυπο το οποίο έχει διανεμηθεί. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο μιλητή να σας πω ότι υπάρχει συνεδρίαση σκιωδών στην ASP 5G3 65 στις 2 η ώρα. Ξεκινάει το απόγευμα. οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες θα παρίστανται. Μπορείτε να θέσετε εκεί τι ερωτήσεις σας και να λάβετε απαντήσεις σε αυτή τη συνεδρίαση, εφόσον η δική μας θα πρέπει να λήξει συντομότατα. Είπαν ότι θα, θα παραστούν εκεί και θα προσπαθήσουν να απαντήσουν τούτων λεχθέντων. Ο λόγος του τελευταίου μιλήτη της συνεδριάσεω αυτή. η κυρία Λανβός από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ. Η, δίκευση, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Έχει το λόγο για σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τι έκανα εγώ σε αυτή την ανάλυση. Βασίστηκα στην κοινή προσέγγιση για όλους τους ε, ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εγκρίθηκε το 2013 από τα τρία θεσμικά όργανα και συγκριτικά στοιχεία. Σύντομα θα κάνω μια παρουσίαση να επικεντρωθώ σε ένα θέμα, στο όνομα και το ρόλο των ενδιαφερομένων κύκλων. Και μετά θα σας περιγράψω τις υφιστάμενες δομές και με ποιον τρόπο η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, θα βασιστεί σε όλη αυτή τη δομή. Για το όνομα, το είπε και ο κύριος Λένας. Για ποιο λόγο αρχή ρωτήσατε. Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ που τη θέσατε. Στην κοινή προσέγγιση το 2012 ορίζεται ρητά και έχει συμφωνηθεί ότι οι μελλοντικοί οργανισμοί θα ονομάζονται οργανισμοί. Οπότε σου λέει γιατί αρχή, γιατί όχι agency και ε, πλέον authority. Θα θέλατε κι εσείς να αναφέρετε ως οργανισμός. Αν δούμε όμως την κοινή προσέγγιση και τις συμφωνίες που έχουν γίνει κανονικά θα έπρεπε να αποκαλείται agency, οργανισμός και όχι αρχή εργασίας. Αυτά ως προς το ιστορικό για να σας θυμίσω κάτι στο οποίο έχετε και εσείς συμφωνήσει. Δεν θα επεκταθώ σε αυτή τη διαφάνεια ε, και σε αυτό το θέμα ε, με χαρά να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ποιο είναι το ιδιαίτερο τώρα σε σχέση με αυτόν τον οργανισμό. Ε, είναι ο ρόλος των ενδιαφερομένων. Ορισμένοι οργανισμοί βάζουν αυτούς τους ενδιαφερομένους στο Διοικητικό Συμβούλιο και ορισμένοι άλλοι δημιουργούν ένα όργανο ad hoc στο εσωτερικό του οργανισμού που είναι και δεν είναι τμήμα του οργανισμού. Στην περίπτωση εδώ της ΕΛΑ, της αρχής εργασίας, έχει το ενδιαφέρον γιατί οι ομάδες των ε, ενδιαφερομένων όπου συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, η ομάδα αυτή εντάσσεται, είναι όργανο του ίδιου του οργανισμού της αρχής αυτής. Αυτό έχει το ενδιαφέρον του σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς. Και από αυτή την προοπτική και τη σκοπιά θέλω να πω κάτι που ανέφερε και ο κύριος Πυρίνσκι για τη σύνθεση. Θέλουμε να συμμετέχουν σε αυτή την ομάδα ενδιαφερομένων και άλλοι. Γιατί στο Διοικητικό Συμβούλιο έχετε τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή των Ενδιαφερομένων Κύκλων έχετε τους κοινωνικούς εταίρους, άρα χάνεται η κλασική τριμερής εκπροσώπηση εργαζόμενοι εργοδότες και ε, κράτος. Κυβέρνηση. Αν παραμείνει αυτή η δομή όμως των ενδιαφερομένων, σε ξεχωριστή επιτροπή, ενδεχομένω θα πρέπει να συμμετέχει εκεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέτε. Που εγώ δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έχει ρόλο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπείται. Πρέπει να συμφωνηθούν θέματα όπως ποιος θα προεδρεύει, πού θα συνεδριάζουν και πότε. Σε άλλους οργανισμούς ή ομάδες ενδιαφερομένων λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Συγκαλούνται μεταξύ τους, προεδρεύουν κάποιος από την ομάδα. Στη γραπτή μου πρόταση έχω κάνει κάποιες προτάσεις αλλαγής αυτών. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω έχει να κάνει με τις υφιστάμενες νομές και πώς θα τις αντικαθαστήσει είναι διάφορες τεχνικές ε, επιτροπές για τη μετακίνηση των εργαζομένων, για την απόσπαση των εργαζομένων, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ε, για την Αδήλωτη Εργασία και ε, ο συντονισμό για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και όπως είπατε θα μπει και το EURES εκεί και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Συντονισμού που εδρεύει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό όλα θα τα αντικαταστήσει η ΕΛΑ. Αυτό που θα συνεχίσει να ισχύει είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή για το Συντονισμό των Κοινωνικών Συστημάτων, η ε, Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ελεύθερη Κυκλοφορία, διάφορα όργανα που είναι ήδη συντεταγμένα και επιτροπές και μια άλλη επιτροπή που μάλλον θα τερματιστεί και θα αντικατασταθεί Οπότε το τελικό κατασκεύασμα θα είναι όπως βλέπετε. Και ποια είναι η προστιθέμενη αξία της ΕΛΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, απλούστευση, απλοποίηση της δομής που υπάρχει τώρα, που έχει όλα αυτά τα όργανα που βλέπετε στη διαφάνεια και θα απομείνουν αυτά, τα τέσσερα. Χωρίς να είναι σαφές σε ποιο βαθμό η ΕΛΑ θα διασυνδέεται με τις υφιστάμενες δομές. Γιατί υπάρχουν κάποιες ε, αρμοδιότητες και κάποια αντικείμενα με επικαλύψεις και δεν τα ξεκαθαρίζει η πρόταση. Συμπέρασμα. Με βάση την ανάλυση μου διαπιστώνω ότι χρειάζεται απλοποίηση και του ρόλου και των αρμοδιοτήτων με συγκεκριμένη αναφορά και απλοποίηση της ε, θεσμικής δομής. Η ΕΛΑ, η ΕΛΕΙ θα βοηθήσει στην απλοποίηση αυτού του, του, του εγχειρήματος της αρχιτεκτονικής, αλλά δεν αρκεί αυτό. With the administrative commission mm. um, Τώρα λοιπόν μήπως έχει έρθει η ώρα να υπάρχουν πιο βαθιές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Το απόγευμα θα τα πει αυτά ο συναδελφός μου στις συνεδρίες. Εγώ δεν τα ξέρω όλα αυτά τα, ε, το εργατικό δίκαιο, δεν είμαι ειδική. Αλλά υπάρχει μια επιτροπή που λειτουργεί πάρα πολύ καλά και δεν θέλει κανείς να τη διαλύσει, ούτε καν να τη θίξει. Αλλά μήπως έχει έρθει η ώρα να αναθεωρήσουμε έτσι πιο ριζικά να γίνει πιο βαθιά μεταρρύθμιση για να υπάρχει μια δομή συνεκτική και λειτουργούσα η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα είναι η ανώτερη αρχή χωρίς να καταργεί, να αντικαθιστά άλλα όργανα. Και μετά θα πρέπει να δούμε ποια σχέση θα διαμορφωθεί ανάμεσα σε αυτή την αρχή και τα κράτη-μέλη. Η Διαχειριστική Επιτροπή όμως, η Διοικητική Επιτροπή ενδεχομένως να γίνει ένα όργανο ευρύτερο ή οργανισμός η ίδια. Αυτή τη στιγμή είναι παράρτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά μπορεί και αυτό να χρειάζεται αναθεώρηση. Ή να περιοριστεί η εντολή της Ευρωπαϊκής να χρειαζεται αναθεωρηση ειναι ειναι περιοριστει Εργασίας που να είναι μόνο αρχή επιθεωρήσεων και επιβολής της νομοθεσίας. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ευρύτερη εντολή τη από αυτό που είχε στο μυαλό του ο κύριο Ιούγκερ όταν ε, τον ανέφερε στην ομιλία του. Άρα και αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί, αν θα έχει ένα ευρύτερο ρόλο ή μόνο τις επιθεωρήσεις και την επιβολή του νόμου και μέχρι εκεί και τα υπόλοιπα εργασιακά αλλού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για τις σύντομες αυτές εκδοχές των παρουσιάσεων. Τα καταφέρατε νομίζω πολύ καλά. Ζητώ συγγνώμη για τη χρονική πίεση. Επαναλαμβάνω ότι όλοι σας είσαστε προσκεκλημένοι, όχι μόνο τα μέλη του Κοινοβουλίου ή τα μέλη της Επιτροπής, τη συνεδρίαση που ξεκινά στις 2 η ώρα στην ASP 5G365 διότι θα είστε εκεί και σε πιο προσωπικό επίπεδο και χωρίς στρες να απαντήσετε σε ερωτήσεις και να δώσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο σας και τις αναλύσεις σας. Σας ευχαριστούμε όλους. Κάνετε κάτι πολύ καλό και χρήσιμο. Σε αυτό το σημείο στη διάταξη. Επόμενη συνέντευξη 7 Ιουνίου, από 9 μέχρι 12.30. Σας ευχαριστώ. Γεια σας και καλό απόγευμα.